Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Γιατί ο υπουργό είναι υπουργό εξωτερικών υποθέσεων και έχει και άλλες ε, αρμοδιότητες ε, και παρουσία σε άλλες επιτροπές. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε για να τον αφήσουμε να συνεχίσει το έργο του και σε άλλες επιτροπές. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Σβέν Μίξερ που είναι ο Εστονός Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και θα συζητήσουμε τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα με ανθρωπιστικές κρίσεις ακόμη και στο κατόφλι μας και στην Μέση Ανατολή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη. Σήμερα το πρωί, κύριε Υπουργέ, συζητούσαμε την κατάσταση στην Ελλάδα, όπου ευτυχώς έχουμε φτάσει από κατάσταση κρίσης σε κατάσταση διαχείρισης ε, μετά την ε, κρίση με τους πρόσφυγες στα νησιά και στην Υπηρετική Ελλάδα, αλλά και στις νότιες ακτές της Ιταλίας ε, έχουμε νέα κρίση τώρα. Κρίσης στην Αφρική, με κατάσταση λοιμού, η κρίση στην Ιεμένη, πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά θα σας δώσω το λόγο και στη συνέχεια σίγουρα θα έχουν ερωτήσει οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που εκφράσατε το ενδιαφέρον σας για τις προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω διότι μου δόθηκε ευκαιρία να συναντηθούμε και το Μάρτιο σε μια προηγούμενη επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες. Ήταν μια συνάντηση πάρα πολύ χρήσιμη για να διαμορφώσουμε το θεματολόγιο της Προεδρίας μας στον τομέα της ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών θεμάτων. Χαίρομαι που σήμερα βρίσκομαι στην Επιτροπή σας για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες της Εστονικής Προεδρίας στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με κάποια μέλη της Επιτροπής σας σε πιο ε, άτυπη συνάντηση σήμερα το πρωί τα θέματα αυτά. Καταρχήν θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της συνεχίζει να είναι ο υπαριθμόν ένα δωρητή ανθρωπιστική βοήθεια στον κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά για την υποστήριξή σα, την δέσμευση που αναλαμβάνετε και την αφοσίωσή σα στα ανθρωπιστικά ζητήματα. Οι ζωντανέ συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ρόλο ελέγχου που έχει το Κοινοβούλιο είναι πολύτιμα. Η ανθρώπινη ζωή έχει ανυπολόγιστη αξία και το να καταστραφεί ακόμη και μία ανθρώπινη ζωή είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό ισχύει σε όλο το φάσμα, από το Ταλίν μέχρι το Χαλέπι. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι θεμελιώδης έκφραση της αποφασιστικότητας του λαού της Ευρώπης να βοηθήσει πολίτες ολόκληρου τον κόσμο που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στην Ευρώπη Ενδιαφερόμαστε και για τους δικούς μας πολίτες, αλλά και για τους πολίτες ολόκληρου του κόσμου, όπου και αν ζουν. Η Εστονία θα βασιστεί στη δυναμική που δημιουργήθηκε από τους συναδέλφους μας από τη Μάλτα και θέλω να ευχαριστήσω την Προεδρία της Μάλτας για το εξαίρετο έργο της όσον αφορά το, την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως πρώτη Προεδρία των, της νέας ομάδας των τριών για τους επόμενους έξι μήνες η Εστονία θα συνεχίσει να προωθεί το συντονισμό για να υποστηρίζουμε μια συλλογική απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στις ανθρωπιστικές κρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι ο αριθμός ε, των παρατεταμένων κρίσεων ε, και το μέγεθος ε, του εκτοπισμού πληθυσμών καθώς και η ανασφάλεια όσον αφορά ε, την ε, διατροφή έχουν φτάσει σε ε, καταστάσεις χωρίς προηγούμενο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Μας ανησυχεί η ανερχόμενη τάση εκτοπισμού πληθυσμών σε περιοχές όπως η Νιγηρία, το Νότιο Σουδάν, η Συρία, το Ιράκ, η Εμένη και άλλες. Και ακόμη και πιο κοντά σε εμά έχουμε ανθρωπιστικές κρίσεις ε, λόγω σειράξεων, όπως στην περιοχή της Ουκρανίας, παραδείγματος χάρη, όπου εκατομμύρια πολιτών αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο Νέλσον Μαντέλα είχε πει ότι πάντοτε φαίνονται αδύνατο να γίνουν τα πράγματα μέχρι τη στιγμή που τα καταφέρνουμε να τα επιτύχουμε. Στον 21ο αιώνα έχουμε τη γνώση, έχουμε τους πόρους και δεν έχουμε δικαιολογία για το να αφήνουμε ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα ή από ανίατες ασθένειες οι οποίες τώρα πλέον έχουν δυνατότητα να ιαθούν. Παρ' όλα αυτά, οι σειράξεις αυξάνουν, γίνονται πιο σοβαρές και καταλήγουν σε ακόμη μεγαλύτερες και πιο επίγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες. Πάνω από 65 εκατομμύρια άτομα έχουν εκτοπιστεί λόγω σειράξεων βίας και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικές καταστροφές, κυρίως λόγω κλιματικής αλλαγής και αύξησης του πληθυσμού, αυξάνονται και γίνονται πιο έντονες. 130 εκατομμύρια άτομα βασίζονται στην ανθρωπιστική βοήθεια σήμερα. Παρ' όλα αυτά, το έργο αυτό δεν είναι αδύνατο να επιτευχθεί και πρέπει να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Η έκθεση τη ε, Επιτροπή Ανατάτου Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών ε, για τη χρηματοδότηση τη ανθρωπιστική βοήθεια τον Ιανουάριο του 2016 Εκτιμά ότι 15 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το έλλειμμα της χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική δράση σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν έχει ακόμη γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Και πιο πρόσφατα, το Μάρτιο του 2017, ο συντονιστής ε, για την ε, βοήθεια επίγουσας ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι σε τέσσερις χώρες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ε, του λοιμού εάν δεν δράσει γρήγορα η παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι λοιπόν το γενικότερο πλαίσιο της κρίσης σε πολλές περιοχές. Το έργο των ανθρωπιστικών φορέων είναι τώρα περισσότερο απαραίτητο από ότι ποτέ. Όσοι δουλεύουν για ανθρωπιστικούς οργανισμούς επισκέπτονται περιοχές όπου υπάρχουν σειράξεις ή καταστροφές για να βοηθήσουν άλλους. Αφήνουν τα σπίτια τους και την οικογένειά τους και οι ίδιοι μερικές φορές έχουν χάσει μέλη της δικής τους οικογένειας είναι θαραλέοι άνθρωποι που αξίζουν το σεβασμό μας και την υποστήριξή μας. Η προστασία των πολιτών είναι βασικός σκοπός κάθε ανθρωπιστικής δράσης. Το να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια σε περιπτώσεις καταστροφής είναι ανθρωπιστική αναγκαιότητα. Αν θυμηθούμε τις ομότητες που διαπράξαν στη Συρία τα τελευταία χρόνια, όπου άμαχοι πολίτες ε, έγιναν στόχος και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεξήχθησαν από αυτούς που πίστευαν ότι μπορούν να παραμείνουν ατιμόρυτοι και αυτό είναι κατάσταση που δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Η Εσθονία ανησυχεί για την μειούμενη ανθρωπιστική υποστήριξη και την έλλειψη πρόσβασης σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε ως κάτι το φυσιολογικό, ούτε ως στρατηγική πολέμου και τονίζουμε την ανάγκη ε, να καταδικάσουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συστηματικά. Η ενεργός επιδίωξη της ανθρωπιστικής βοήθειας με βάση τις ανάγκες και τις προστασίες του ανθρωπιστικού χώρου θα παραμείνει προτεραιότητα για την Προεδρία της Εσθονίας. Δεύτερον, η Προεδρία της Εσθονίας θα αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στις παρατεταμένες εκτοπίσεις ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει το υψηλότερο επίπεδο εκτοπισμού πληθυσμών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό δημιουργεί την ανάγκη να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ανθρώπων που πλήττονται μακροπρόθεσμα. Τα τελευταία 15 χρόνια ο αριθμός προσφύγων και μεταναστών σε ολόκληρο τον κόσμο μεγαλώνει περισσότερο από τον ε, παγκόσμιο πληθυσμό. Οι κρίσεις σήμερα, είτε φυσικές καταστροφές είτε ανθρωπογενείς καταστροφές, δεν μπορούν να επιληθούν μόνο με ανθρωπιστικά μέσα. Πρέπει να συγκεντρώσουμε την πολιτική μας βούληση και το θάρρος μας, να σταματήσουμε και να ανατρέψουμε αυτή την ζωφερή τάση και να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε που αποτελούν τη ρίζα της. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των χωρών που είναι εταίροι μας για να εμποδίσουμε τις, να προλαμβάνουμε τις κρίσεις και η έννοια της ανθεκτικότητας έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Από ανθρωπιστική προοπτική δεν έχει αλλάξει πολύ, αλλά η ενίσχυση της ανθεκτικότητας είναι ουσιώδης για να μπορέσουν οι ευάλωτες χώρες να γίνουν περισσότερο ανθεκτικές και να εξαρτώνται λιγότερο στην εξωτερική βοήθεια και παραμένει στην καρδιά των προσπαθειών μας το να μειώσουμε τις ανθρωπιστικές ανάγκες, να σώσουμε ζωές και να αποφύγουμε την ταλαιπωρία των πολιτών. Χαιρετίζουμε λοιπόν τη νέα στρατηγική προσέγγιση ως προς την ανθεκτικότητα. Η νέα στρατηγική της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει τη σημασία του να βοηθούμε χώρες, κοινωνίες, κοινότητες και άτομα να προσαρμοστούν στις αυξανόμενες πιέσεις ε, που δημιουργούν σειράξεις και χαιρετίζουμε τη στενή συνεργασία των φορέων σε ευρωπαϊκό, ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο, τηρώντας ε, τις εντολές ε, που έχουν δοθεί και τις ανθρωπιστικές αρχές. Προετοιμαζόμενοι για τις δράσεις ε, και ανταποκρινόμενοι σε κρίσεις, υποστηρίζουμε ένα ισχυρότερο ανθρωπιστικό πλαίσιο ε, σε δίκτυο με την ανάπτυξη. Όπως ε, δήλωσε η Νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη, η φτώχεια, οι συγκρούσεις, ο ευάλωτος χαρακτήρας και οι εκτοπισμοί πληθυσμών συσχετίζονται άμεσα και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο οι θετικές συνέργειες ε, μπορούν να βοηθήσουν. Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε για να διασφαλίσουμε πιο στενή συνεργασία μεταξύ των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών φορέων, καθώς και αυξημένη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που περιλαμβάνουν και διμερείς κρατικούς οργανισμούς και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και την κοινωνία των πολιτών και τις ε, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης. Πρέπει όλοι να εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουμε την ε, συνεισφορά μας στη συμπληρωματικότητα και στη συνοχή της διεθνούς υποστήριξης σε λαούς που υποφέρουν σε ευάλωτες καταστάσεις που πλήττονται από συγκρούσεις. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουμε για την ανθεκτικότητα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε τους πληθυσμούς ε, που πλήττονται από τις συγκρούσεις και τις κρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Προωθούμε την υποστήριξη των παιδιών και των νέων, οι οποίοι είναι φυγάδες από καταστάσεις πολέμου, ιδίως προωθούμε την πρόσβασή τους σε ασφαλές περιβάλλον ποιοτική εκπαίδευσης, καθώς και σε υπηρεσίες προστασίας. Και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους πολίτες. Ε, τρίτο σημείο, η Εστονική Προεδρία παραμένει ισχυρά δεσμευμένη στην υποστήριξη της ε, του φιλόδοξου ανθρωπιστικού θεματολογίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και των βασικών δεσμεύσεων, όπως εγκρίθηκαν στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη κορυφή πέρυσι στη Κωνσταντινούπολη. Η Διάσκεψη κορυφή ζήτησε να υπάρξει μια αλλαγή στην ανθρωπιστική δράση. Ανελήφθησαν σημαντικέ δεσμεύσει για την πρόληψη των συγκρούσεων και του εκτοπισμού. Στο πνεύμα λοιπόν αυτής της παγκόσμιας ανθρωπιστικής διάσκεψης, η Εσθονία θα εστιάσει στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας και στην καινοτομία για τις ανθρωπιστικές λύσεις. Η Μεγάλη Συμφωνία, η αποκαλούμενη Grand Bargain, είναι μια διαδικασία που δημιουργήθηκε μετά ε, το, την Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρωπιστική Χρηματοδότηση και είναι μία από τι λύσει για να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα τη χρηματοδότηση. Ε, είναι πραγματικά μια συμφωνία μεταξύ των δωρητών και των χωρών που κάνουν την υλοποίηση και απαιτεί εμπιστοσύνη από όλε τι πλευρέ. Η Ιστονική Προεδρία υποστηρίζει τι πιο αποτελεσματικέ πρακτικέ μεταξύ δωρητών και ε, ε, οργανισμών που παρέχουν βοήθεια. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν και αύξηση της ευελιξίας στη χρηματοδότηση, περισσότερο πολιετής συνεισφορές, προγραμματισμό των πληρωμών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης. Ζητούμε από όλου του εταίρου να συμφωνήσουν με τη διαδικασία τη μεγάλη συμφωνία που θα αποτελέσει εργαλείο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη ανθρωπιστική βοήθεια, διαφάνεια και εμπιστοσύνη. Οι ανθρωπιστικοί φορεί αναμένεται με λιγότερα μέσα να επιτύχουν περισσότερα και οι νέε προκλήσει δημιουργούν νέε προσεγγίσεις. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα για να έχουμε θετική επίπτωση στην ανθρωπιστική διαδικασία. Θέλουμε και ο ιδιωτικός τομέας να βοηθήσει στην ανθρωπιστική βοήθεια για να, για να μεγιστοποιήσουμε την καινοτομία, να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για να έχουμε πιο απλές και λιγότερο κοστοβόρες λύσεις, με τρόπο πιο αποτελεσματικό και διαφανή. Απευθυνόμενοι σε νέους εταίρους, θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουμε εστιασμένοι στις βασικές ανθρωπιστικές μας αξίες. Παράλληλα με τη συνέχιση που δίδεται στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφή, η Εστονική Προεδρία θα διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια θα λειτουργήσει ω βασικό στοιχείο αναφορά για τα κράτη-μέλη και την ανθρωπιστική του δράση και ιδίω στο πλαίσιο τη δεκάτη επαιτίου τη συνένεση το Δεκέμβριο του 2017. Θέλουμε να δούμε ε, πρόοδο και στην ε, μείωση της βίας ε, βάσει του φύλου. Η συμμεταχείριση των γυναικών και ανδρών θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την εξάλληψη της φτώχειας και αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να ισχύσει και σε περιοχές σειράξεων. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έχουν σχέση με το φύλο και στα ανθρωπιστικά και αναπτυξικά μας προγράμματα. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις γυναίκες ως φορείς αλλαγής στην ανθρωπιστική ε, ανταπόκριση, ούτως ώστε οι λύσεις να είναι σωστά σχεδιασμένες και να συμπεριλαμβάνουν τις γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το να έχουν ε, Λόγω, οι γυναίκες επιτόπου σε περιοχές που πλήττονται από την κρίση θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το υψηλό επίπεδο βίας βάση του φύλου σε καταστάσεις όπου οι γυναίκες και τα παιδιά περιθωριοποιούνται και είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες της Ιστονική Προεδρίας για το ανθρωπιστικό πρόγραμμα και η φιλοδοξία μας είναι να συνεργαστούμε μαζί σας για να προωθήσουμε πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και να αντιστρέψουμε την αρνητική ε, αυξητική, την αρνητική ε, κατάσταση όπου αυξάνεται, αυξάνονται οι τοπισμοί και θέλουμε να δημιουργήσουμε καινοτόμες ανθρωπιστικές λύσεις. Προβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επισκόπηση. Σίγουρα οι συνάδελφοι έχουν διάφορες ερωτήσεις. Να δώσω πρώτα το λόγο στον Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παραθέσατε τις προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας. Το βέβαιο είναι ότι συχνά συμβαίνει το εξής. Οι κατάλογοι προτεραιοτήτων των Προεδριών να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, τα προβλήματα δεν λύνονται μόνο εντός εξαμήνου, παραμένουν, επιλύονται σε βάθος χρόνου και είναι λογικό η επόμενη Προεδρία να θέτει ως προτεραιότητες ε, αυτές που είναι αρκετά κοντινές ε, με τις προτεραιότητες της προηγούμενης Προεδρίας. Και πιστεύω ότι και αυτά θα απασχολήσουν την επόμενη από εσάς Προεδρία, την Βουλγαρική Προεδρία. Από την παρέμβασή σας βεβαίως ε, κρατάω ότι υπάρχει συμφωνία. Πράγματι, αυτές είναι οι προτεραιότητες με τις οποίες πρέπει κανείς να ασχοληθεί κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και συμφωνώ μαζί σας. Έχω κάποια σχόλια να κάνω και κάτι να σας ζητήσω, κάτι να σας ρωτήσω. Κάποια στιγμή Μιλήσατε για την αντοχή, για την αθεκτικότητα και είπατε ότι η άποψη για όλα αυτά έχει προχωρήσει, έχει κερδίσει έδαφος σε όλο αυτό το πεδίο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, όμως έχει κερδίσει λιγότερο έδαφος ε, ό,τι έχει να κάνει με την ανθρωπιστική βοήθεια ή ανθρωπιστική δράση. Όμως και ωστόσο και ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων όπως και με το ότι έχει να κάνει με την πρόληψη και ανταπόκριση και αντίδραση σε καταστροφές φυσικές. Η ανθεκτικότητα, η αντοχή είναι καθοριστικό στοιχείο σε αμφότερα τα πεδία. Ερχόμαστε από μια διάσκεψη των ΗΠΑ στην Κανκούν για τη μείωση των κινδύνων για την έλευση φυσικών καταστροφών σε περίπτωση που σημειώνονται τέτοιου είδου φυσικές καταστροφές. Περισσότερε λεπτομέρειε θα σα πω κάποια άλλη στιγμή. Ε, μετά από τις συμφωνίες του, Σεντάι και μετά από δύο χρόνια μετά από αυτές τις συμφωνίες, κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση αξιολόγηση δόθηκε έμφαση πάλι στο σκέλος της προετοιμασίας, της πρόληψης, της ε, Προσπάθεια ύπαρξης μιας στρατηγικής αθεκτικότητας, αντοχής, αντίστασης όταν σημειώνονται τέτοιου είδους καταστροφές. Τα στοιχεία δεν λένε ψέματα. Σώνονται πολύ περισσότερες ανθρώπινες ζωές, εξοικονομούνται πολύ περισσότεροι πόροι εάν οι κοινωνίες είναι καλύτερα προετοιμασμένες και είναι σε θέση να ανταποκριθούν, να απαντήσουν με αποτελεσματικότητα σε τέτοιου είδους ενδεχόμενα. Αυτό καταρχάς. Το δεύτερο που κρατώ από την παρέμβασή σας είναι κάτι που ενδιαφέρει τα μάλα την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Ανάπτυξης. Δηλαδή θέλουμε την ανθρωπιστική βοήθεια να τη συνδέσουμε με την ανάπτυξη επιτόπου. Ο σύνδεσμος, ο κρίκος που θα συνδέει την ανθρωπιστική βοήθεια με την αναπτυξιακή δραστηριότητα είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η ανθρωπιστική απάντηση επέρχεται σε επίγουσες και κατεξαίρεση συνθήκες, αλλά θα πρέπει να ριζώσει για να μετατραπεί σιγά σιγά σε αναπτυξιακή βοήθεια και όσοι δέχονται τις πρώτες βοήθειες να μπορέσουν να μετατρέψουν αυτή τη στήριξη σε στήριξη για την ανάπτυξη και την πρόοδό τους. Υπό αυτή την έννοια, η παρακολούθηση της Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη ε, είναι κάτι το σημαντικό και λογικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το εξάμεινο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες του χρόνου να μας παρουσιάσει έναν απολογισμό για το πώς δρομολογήθηκαν οι δεσμεύσεις που προσυπογράφτηκαν στην Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής της Κωνσταντινούπολης και από πλευράς της Ένωσης των νομικός φορέας και διεθνής φορέας και από πλευράς των κρατών μελών. Χρειάζεται όθηση από το Συμβούλιο έτσι ώστε οι χώρες μέλη να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο θα έλεγα. Και αυτό το στοιχείο θα πρέπει να συνοδεύει τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διάφορες δεσμεύσεις και για το σχέδιο δράσης. Προς το τέλος της παρέμβασής σας νομίζω ότι αναφερθήκατε σε κάτι σημαντικό. Η καινοτομία ήταν ένα από τα στοιχεία κλειδιά στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, ό,τι έχει να κάνει με την ανθρωπιστική βοήθεια. Μιλούμε για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, νέους μηχανισμούς, νέες απαντήσεις. Τον ε, Σεπτέμβριο, ως εκ τούτου, θα αναλάβει δραστηριότητα η δική μας Επιτροπή σε ό,τι έχει να κάνει με το πεδίο της καινοτομίας στην ανθρωπιστική βοήθεια και θα παρουσιαστεί μια μελέτη την οποία εμείς ως Επιτροπή έχουμε αναθέσει, έχουμε αναθέσει την εκπόνησή της δηλαδή και θεωρώ ότι η Προεδρία πρέπει να δράξει αυτή την ευκαιρία για να δούμε που βρισκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με την καινοτομία στο πεδίο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και ως προς τα δύο τελευταία σημεία γίνεται συζήτηση το κατά πόσο 10 χρόνια μετά την έγκριση της υφιστάμενης συνένεσης αξίζει να αναθεωρηθεί και να μεταρρυθμιστεί το πλαίσιο αυτής της συνένεσης. Θα άξιζε πιστεύω να γίνει μια δημόσια ανοιχτή συζήτηση για το αν είναι επαρκής η συνένεση που διαθέτουμε ή αν χρειάζεται να ε, τα αλλάξουμε αυτά και να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία. Τέλος, Έχω να πω το εξή. Όταν μιλούμε για ανθρωπιστική βοήθεια, κατά κύριο λόγο δεν σκεφτόμαστε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, υπάρχουν καταστάσεις εντό ευρωπαϊκή Ένωσης που απαιτούν να υιοθετήσουμε την οπτική γωνία Τη ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν λέω να υιοθετήσουμε τους πόρους αυτούς κάθε αυτού, αλλά την ερμηνεία, την οπτική γωνία. Και αφού είστε υπεύθυνο στο Συμβούλιο και αρμόδιο για τα θέματα αυτά, σα ζητώ να λάβετε υπόψη σα ότι ό,τι γίνεται για μετανάστες, πρόσφυγες και του των ε, ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να κάνετε προώθηση και προαγωγή της ιδέας ότι και αρμόδια υπουργικά χαρτοφυλάκια που έχουν σχέση, να που έχουν σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια αξίζει να ε, καθίσουν στο τραπέζι ε, και να μην είναι μόνο οι Υπουργοί Εσωτερικών αρμόδιοι για όλα αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ θερμά η Πρόεδρος. Όταν υπήρξε η χρηματοδότηση ΕΚΟ στην Ελλάδα και είχαμε εμπειρογνωμοσύνη για την ανθρωπιστική βοήθεια από πλευρά ανθρωπιστικής βοήθεια, τότε βελτιώθηκαν τα πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει διάφορε κρίσει και ξέρουν ακριβώ τι να κάνουν και πώ να γίνουν γρήγορα όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά συζητήσαμε και σήμερα το πρωί και ίσως κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και συμβαίνει στην Ιταλία. Έχω τέσσερι ομιλητές, Βαντεβέντε, Χόιμπουκ, Λίντς και Σεσίλ Κιέγγε. Τέσσερις έχουν εγγραφεί στο κατάλογο των ομιλητών. Νόρμπερτ και εσύ. Καλώς. Πέντε. Ο κύριος Νόιζερ δηλαδή. Ξεκινάμε με τον κύριο Βέντα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και εσάς κύριε Υπουργέ μας προσιάζετε τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας, λέει ο κύριος Βέντα. Η πρώτη ερώτηση αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια για τον σχεδιασμό της. Δεν θα πρέπει να έχουν κάποιο είδου αξιόπιστη εποπτεία, κάποιο μηχανισμό αναφορών τόσο ώστε να μπορεί η Ένωση και τα κρατημέλη ε, να μπορούν να είναι υπόλογοι για τις ε, υποσχέσεις και δεσμεύσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Επίσης, όπως μας είπατε, προηγουμένως, Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε κάποιο είδου ψηφιακές συσκευέ που να χρησιμοποιούνται για την αναπτυξιακή πολιτική. Τι πιθανότητες υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν αυτές πραγματικά από τα κρατημέλη, γιατί ήταν το θέμα της χρηματοδότησης όπως είπατε και όπως ξέρετε η θέσπιση νέων χρηματοδοτικών μέσων για την ε, σωστή διακυβέρνηση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δημοκρατία, όλα αυτά είναι ε, πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά τι ισχύει στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις που ίσως προχωρούν και λίγο περισσότερο και αφορούν το πρόγραμμα εργασίας της Ιστονίας για την αναπτυξιακή πολιτική που έχει σχέση και με την, το θεματολόγιο του 2030, τις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ και την ανθεκτικότητα. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για την καταπολέμηση των αιτίων της, του εκτοπισμού. Υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα τα οποία πρέπει να γίνουν πιο συνεκτικά και πιο ολοκληρωμένα. Τι θα μπορούσατε να μας προτείνετε σχετικά και πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε, ποια θα είναι τα μέσα με τα οποία θα χειριστείτε αυτή την κατάσταση. Επίσης, όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας, μιλάμε για συνεκτικότητα, αλλά όχι σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική. Και συμπεραίνω ότι για την Εστονική Προεδρία δεν θα αποτελέσει προτεραιότητα αυτό. Μου φαίνεται περίεργο, διότι για την πολιτική ε, της συνοχής δεν υπευλήθησαν ε, εκθέσεις και αν, ε, από πλευράς της Επιτροπής και αν και το Συμβούλιο δεν το θέσει ως προτεραιότητα δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την επίσκεψη στην Επιτροπή μας. Εμείς ευχαριστούμε. Λίζ. Σα άκουσα ε, πάλι ιδιότητα χθε ω Υπουργό Εξωτερικών ότι έχουν συνέπεια αυτά τα οποία μα λέτε και εμεί αλλάζουμε ρόλου τέλο πάντων. Έχουμε επισκεφθεί κάποιοι εξημών χώρα σας και επίσης και εμείς εδώ στις Βρυξέλλες ε, ασχολούμαστε με ανθρωπιστικές κρίσεις και μέρα και νύχτα ασχολούμαστε με τις τραγωδίες όλο τον κόσμο. Πάντως ακόμα ε, δεν υπάρχει κάλυψη των αναγκών από πλευρά νοσοκομείων. Εκεί πάσχει η ευρωπαϊκή προσέγγιση. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο ώρες πάνω σε αυτό. Επίσης από πλευρά σοσιαλδημοκρατών Θα θέλαμε η ανθρωπιστική βοήθεια να αφιερωθεί κατά ένα κομμάτι της στα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης γιατί αυτά τα πράγματα μαθαίνουν οι νέοι. Μήπως θα μπορούσατε να το κοιτάξετε και αυτό. Να καλύψουμε επομένω και τους νέους και τις γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις. Και έτσι να πάμε πέραν των ε, ανηλίκων και στο θέμα της ε, χειραφέτησης μέσα από την παιδεία των γυναικών. Κέγγε. Ευχαριστώ για το πρόγραμμα το οποίο μας παρουσιάσατε. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Πρώτα πρώτα, ασχολούμαι με τις χώρες ΑΚΕ και θα ήθελα πάνω σε αυτά να σας πω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις χώρες ε, ΑΚΕ ε, βλέπω στο πρόγραμμά σας είναι μία προτεραιότητα. Μας μίλησατε για τους νέους και ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα για αυτούς στα πλαίσια της στρατηγικής σας. Επίσης να καλύψετε και τις γυναίκες όπως είπατε στην ομιλία σας. Να δείτε πως θα υπάρξει κάποια ανθεκτικότητα ε, όσον αφορά την κάλυψη νέων και νέων γυναικών. Γιατί πρόκειται για ευπαθή, την κατηγορία. Αλλά αυτό που δεν βρίσκονται στη στρατηγική σα είναι κάτι για την διασπορά. Πρόκειται για εκείνους οι οποίοι πολύ καιρό ζουν εκτός Αφρικής. Εν προκειμένου που ζουν πολύ καιρό στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να γυρίσουν στην Ήπειρο καταγωγής τους. Δεν βλέπω κάποια κάλυψη για εκείνους. Τι θα μπορούσατε να κάνετε για αυτή την κατηγορία. Δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά το έργο σας, την υποστήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας σε κάποιες περιπτώσεις κατεπίγουσες και αναφέρομαι πρώτα-πρώτα για αυτά τα οποία γίνονται στο Κονκό. υπάρχει βοήθεια αλλά υπάρχουν και οι σφαγές. Εσείς θα συνεχίσετε την υποστήριξη των εκεί προγραμμάτων. Επίσης για τις νέες γυναίκες στην Ιγυρία. Γνωρίζω ότι έχουμε αυτές τις νέες, τις 200 κοπέλες που απήχθησαν θύματα της Μπόκο Χάραμ. Θα βρίσκονται στο Καμερούν, στην Ιγυρία, ε, είναι σε πάρα πολύ επικίνδυνη φάση τώρα αυτό το πρόβλημα όπως μάθαμε από λίγες μέρες. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Πολλά μπορούμε να κάνουμε και κυρίω να δούμε τι θα γίνει με τις απότερες αιτίε. Αλλά ό,τι κάνουμε να βρίσκει συνέχεια. Πλούσιο το πρόγραμμα της Προεδρίας σας, αλλά παρακαλώ απαντήστε μου σε αυτά τα ερωτηματάκια. Ευχαριστώ. Εμείς λέει Πρόεδρος ο κύριος Νόιζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι το θέμα της ασφάλειας και της μετανάστευσης καλύπτει όλο και περισσότερο κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μην ξεχνάμε και το βασικό στόχο της Επιτροπής μας, την καταπολέμηση της φτώχειας. Στην διάσκεψη κορυφής, τέλος Νοεμβρίου στην Αθήνα του του, θα είναι ρόλο της δικής σας Προεδρίας να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και σήμερα έχουμε και την έκθεση του συναδέλφου Μωρίς Πόγκα. Πρέπει να δούμε πώ εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να έχουμε καλή συνεργασία με την Αφρική και θα ήθελα να ακούσω ε, από εσά ως Προεδρεύοντα του Συμβουλίου πώς βλέπετε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρική; Συμφωνείτε με τη γνώμη μου ότι η καταπολέμηση της φτώχειας είναι μια προεξάρχουσα αρχή χωρίς βέβαια να παραμελούμε τις νέες προκλήσεις της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Και υπάρχει και το ερώτημα του τι γίνεται για τη συνέχεια του Κοτονού. Ξέρω ότι ορισμένα κράτη-μέλη ε, δυσκολεύονται να καταλάβουν τους διαφορετικούς ε, τρόπους συνεργασίας με την Αφρικανική Ήπειρο ε, και με την Αφρικανική Ένωση. Είναι ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Εστονική Προεδρία καθώς και η Βουλγαρική Προεδρία στη συνέχεια. Θέλουμε να έχουμε ένα καλό μέλλον, μια καλή προοπτική για μετά τη Συμφωνία του Κοτονού. Ιδίω διότι θέλουμε να υπάρχει ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ρωτήσατε πολλά που είναι και εκτό θέματο ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι η τελευταία μα συνάντηση πριν τι θερινέ διακοπέ. Οπότε θα σα τη χαρίσω. Και τέλο πάντων, α απαντήσει ο κύριο Υπουργό σε όποια πρόταση μπορεί. Ξέρω ότι ξέρει πολλά γιατί φάγαμε μαζί και ξέρω ότι έχει ευρύτατε γνώσει. Αλλά έχει δικαίωμα να μα πει ποια προτιμά να απαντήσει και ποια όχι. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε τα ανθρωπιστικά προβλήματα στην Ελλάδα, όπου χρηματοδοτούμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Στην Ιταλία επίσης συνεχίζεται η κρίση. Το Συμβούλιο το συζήτησε. Δεν ξέρω αν έχει ζητήσει και η Ιταλία βοήθεια ε, όπως ε, η Ελλάδα και να δούμε τι θα κάνουν ε, οι Υπουργοί για να αντιμετωπιστεί η κρίση στη Μεσόγειο. Ο υπουργό, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα ρωτήσατε. Κατάλαβα ότι θα επικεντρωνόμασταν στα ανθρωπιστικά. Και τα θέματα τα αναπτυξιακά θα τα συζητούσα μάτυπα πριν τη συνεδρίαση. Γι' αυτό και δεν ε, έφυξα τα θέματα της ανάπτυξης. Επειδή αυτά αφορούν περισσότερο την είπατε εκπρόσωπο και όχι τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Να σας πω τα θέματα τα αναπτυξιακά πάντως τα της ε, νομισιακής βοήθεια και νομισιακής συνεργασία. Να κάνω ό,τι μπορώ να τα πούμε και αυτά. Πρώτα πρώτα. Όσον αφορά αυτά τα οποία ρώτησε ο κύριος Γκερέρο Σαλόν, ναι, σε πολλές περιπτώσεις οι προτεραιότητες δεν αλλάζουν ε, σημαντικά από προεδρία σε προεδρία. Και αυτό για διάφορους λόγους. και παγιώ ε, ασχολούμαστε με κάποια ζητήματα όπως ε, η αντιμετώπιση της ε, φτώχειας, το πώς θα προστατεύσουμε τις πιο ευάλωτε χώρες, Αυτού που είναι οι βασικοί αποδέκτες της ανθρωπιστική βοήθειας. Επίσης, αυτό ισχύει γιατί πολλές από τις κρίσεις παρατείνονται αποτελούν, αποκτούν μάλλον μόνιμο χαρακτήρα. Οπότε θα πρέπει παράλληλα να κάνουμε τουλάχιστον δύο πράγματα. Να ασχολούμεθα με τα πιο κατεπήγοντα, να δίνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που υποφέρουν, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επίλυση πιο μακροπρόθεσμων προβλημάτων. Και κάποια αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράμματα. Θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στο να βρεθεί κάποια βιώσιμη λύση για κάποιες πάγιες μόνιμες ε, κρίσεις. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, θα συνεχίσουν οι κρίσεις και επί Βουλγαριακής και επί Αυστριακής ε, ε, Προεδρίας και στο μέλλον και μετά δηλαδή από αυτές. Δηλαδή είμαι αισιόδοξο, αλλά είμαι και ρεαλιστής γιατί θα πρέπει να δεχθούμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα διαρκέσουν τόσο αφορά την ανθεκτικότητα και για τις φυσικές καταστροφές ε, και για τις καταστροφές που προέρχονται από τον άνθρωπο ε, είναι μια κρίσιμη έννοια. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν τέτοιες δομές ανθεκτικές για τους πιο ευάλωτους. Για τις χώρες και για τους λαούς που επανειλημμένα πλήσονται από τέτοιες καταστροφές. Έτσι εξοικονομούμε και το χρήμα των φορολογουμένων όταν υπάρχουν ε, επιτόπου κάποιες δομές ανθεκτικότητας και αντοχής για αυτές τις χώρες. Και έτσι μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει εκ των υστέρων τις συνέπειες των ε, θεομηνίων. Περισσότερο από τις ε, καθώς από τον άνθρωπο. Συγκρούσεις κλπ. Άρα, αξίζει να ασχοληθεί κανείς με αυτή τη λύση, οπότε και εμείς έχουμε βοηθήσει στο θέμα της ε, ανθεκτικότητας. Και έτσι οι χώρες ε, αποδέκτες να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους κινδύνους κάθε είδους δηλαδή καταστροφή και κρίση. Ερωτήθηκε κάτι για την μετανάστευση και κατά πόσο αυτό θα πρέπει να είναι θέμα υπουργών εσωτερικών. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα αδιέρετο η ασφάλεια μέσα στην παγκοσμιοποίηση που ζούμε. Τι διάκριση να κάνουμε για ε, εσωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική και μετανάστευση για την ε, ε διάφορες μορφές ασφάλειας hard και soft είναι αδιέρετη η ασφάλεια Λέμε για εσωτερικά, εξωτερικά χαρακτηριστικά της μετανάστευσης. Θα πρέπει να συνεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες αρμονικά. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπηρεσίες των χωρών προέλευσης. Όταν μιλούμε για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση και στα σύνορα αυτής, θα πρέπει αυτό να γίνεται, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε αυτών των μεταναστευτικών ροών. Χρειάζεται δηλαδή μια σφαιρική προσέγγιση στο μεταναστευτικό και να δεχθούμε ότι οι λαοί και οι άνθρωποι γενικώ ανέκαθαν μετακινούνται. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε τη μετακίνηση 100%. Υπάρχει και η διάκριση λάθρο μετανάστευσης και νόμιμης μετανάστευσης. Οπότε θα πρέπει να είναι δυνατόν κάποιος όταν δικαιούται να μετακινείται όταν έχει αντιμετωπίσει μια ε, καταστροφή, κάποια σύγκρουση ή όταν ε, αναζητεί μια καλύτερη ζωή για αυτόν και τα παιδιά του. Τώρα για τον κύριο Βέντα όσον αφορά ε, τους ενωτησιακούς στόχους SDGs, το θέμα της απόδοση ευθυνών και της λογοδοσίας, τα είπαμε στο γεύμα Είπαμε ότι θα πρέπει ε, να θέσουμε στόχους, τους οποίους να επιδιώξουμε σε σχέση με τους πόρους που διαθέτουμε σαν τεξιακή συνεργασία ή στην ανθρωπιστική βοήθεια. Και συγκεκριμένα για συγκεκριμένα προγράμματα και μέσα. Είναι θλιβερό όταν κανείς δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους που ο ίδιος έταξε. Ε, δεν υπάρχουν ε, δικαιολογίε όταν κανείς δεν τα καταφέρνει σε αυτό το επίπεδο. Λίγα χρόνια μένουν για τον στόχο του 2030. Πλησιάζουμε το ορόσημο κοινό. Όλο ένα και περισσότερο φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουν όλοι να πετύχουν τους σχετικούς στόχους. Ε, βέβαια, είναι κάτι το απαιτητικό από πολιτικής πλευράς το να πετύχεις τους στόχους. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα χρήματα τα οποία έχουμε ως κρατή-μέλη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδέψει στα ανθρωπιστικά είναι όλο ένα και περισσότερα. Αλλά δεν μπορέσαμε να συμβαδίσουμε με την ανάγκη που υπάρχει. Και να αυξήσουμε αυτά που διαθέτουμε όταν έχουμε κάποιου είδου ε, θεομηνίες και καταστροφές. Τώρα χρήση ψηφιακής τεχνολογίας από τα κρατημέλη. Οι ψηφιακές λύσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένας καλός τρόπος να υπάρχει περισσότερη εργοδοσία, περισσότερη διαφάνεια και επιταχύνει κιόλας την ε, παροχή της βοήθειας. Συμφωνούμε σε αυτό, όμως είναι το θέμα της γνώσης των ψηφιακών. Και βέβαια, σε σχέση με το ποιος θα παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, Υπάρχουν διαφοροποιήσει από χώρα σε χώρα. Πάντω εν γέννη, υπάρχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Άρα θα πρέπει να πασχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση. ούτως ώστε να αποκτήσει περιεχόμενο αυτή η ιδέα, αυτή η έννοια. είναι καινοτόμος μέθοδος αντιμετώπισης και επίτευξης των στρατηγικών στόχων. Και πολλές από τις φτωχές χώρες θα συνεχίσουν να έχουν παραδοσιακές οικονομίες για πολλά χρόνια. και χρειάζονται υποδομές για να μπορέσουν να πούμε να μεταφέρουν τα προσεμπορία αγαθά τους και θα ενεργούν παραδοσιακούς τρόπους σε σχέση με την ευρωπαϊκή βοήθεια. Πάντως όμως μπορούμε, γιατί να μην μετέλθουμε και αυτό το μέσο της ψυχικής τεχνολογίας. Τώρα, άλλη ερώτηση. Κύριε Χόιμπουχ, καταπολέμηση των αιτιών της μετανάστευσης με τρόπο συμπληρωματικό και συνεκτικό. Ε, βέβαια, όπως προείπα, Πώς να φρενάρουμε 100% τη μετανάστευση. Θα πρέπει να δούμε βέβαια τις αιτίε γιατί αναγκάζει το κόσμος να μεταναστεύσει. Γιατί θα πρέπει να διακινδυνεύει με τέτοια ταξίδια, γιατί θα πρέπει να πληρώνει εγκληματίες για να ξεφύγει από εμφυλίους και από καταστροφές. Βέβαια, τις ρίζες του φαινομένου θα πρέπει να τις ε, χειριστούμε, αντιμετωπίσουμε με τρόπο βιώσιμο. Έχουμε μια όρημη προσέγγιση και συνεργασία, όπως προανέφερα. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη είναι προτεραιότητα για την Προεδρία μας στο ίδιο επίπεδο με την ανθρωπιστική βοήθεια. Αφήστε που θεωρώ ότι αυτά πάνε χέρι-χέρι, αυτές οι πολιτικές. Γιατί μακροπρόθεσμα έχουν την ίδια κατάληξη, δηλαδή το πώς θα θωρακιστεί μια κοινωνία, τόσο ώστε να είναι σε θέση να προστατευτεί, να αντέξει σε πιέσεις έντονες, να μπορεί μια κοινωνία να κινητοποιηθεί και σε σχέση με θεομηνίες και άλλου είδους κρίσεις. Πάντως σας πω την αλήθεια, θεώρησα ότι σήμερα θα συζητήσουμε κυρίως τα της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας και όχι τόσο τα της ε, ανάπτυξης, που πάντως σημαίνει προτεραιότητα για την ε, ε, Προεδρία μας. Τώρα για τον κύριο Λίτς. Έλλειψη νοσοκομείων. Και ανθρωπιστική βοήθεια που να πηγαίνει και στην παιδεία. Ε, βέβαια και η ιατρική ε, κάλυψη χρειάζεται. Ε, βέβαια και θα το προσέξουμε. Να υπάρχουν ιατρικές υπηρεσίες ποιοτικές. Τώρα όσον αφορά την παιδεία. Είναι σημαντικό στοιχείο της ε, ανθρωπιστικής μας προσπάθειας αλλά και της ε, πολιτικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην παιδεία σε περιοχές και σε χώρες όπου σοβούν οι κρίσεις. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος ούτως ώστε να καταπονήσουμε τη φτώχεια, να δώσουμε κάποια ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα στις ε, χώρες αυτές και Επίσης, έτσι θα καλύψουμε και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γυναίκες, μειονότητες. Είναι κάτι εξοχήν, μια δόκιμη στρατηγική, πρόσβαση στην παιδεία, βελτίωση αυτής. Και συνοδευτικά να δίνονται ευκαιρίες πρόσβαση δηλαδή στην αγορά και ευκαιρίες οικονομικού χαρακτήρα για τους νέους. Είναι πολυδιάστατο πρόβλημα αυτό και πρόκληση. Τώρα, δεν ξέρω το όνομά σας, πώς προφέρετε, κυρία Κίνγκα. Ελπίζω δεν Έκανα και πολύ μεγάλο λάθος την προφορά. Για την Αφρική. Και τα θέματα της διασποράς. Ε, βέβαια. Είναι σημαντικό το θέμα. Ναι, δεν το ανέφερα, αλλά είναι στο θεματολογιό μας και θα λάβω υπόψη αυτό το οποίο είπατε. ευχαριστω είναι Να λεφτεί υπόψη αυτό που είπατε. Είναι σημαντική προτεραιότητα επίσης η Αφρική. και σε σχέση με την συνάντηση κορυφής Ευρώπη Αφρική τον Νοέμβριο στο Αμπιτζάν όπου θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις συνεργασίας με την Αφρικανική Ένωση με τις Αφρικανικές χώρες την Αφρικανική Ήπειρο και έχουμε το θεματολόγιο του 2063 έχουμε τον προγραμματισμό στρατηγικής πολιτικής που ενσωματωνόνται σε διαφορά έγγραφα, οπότε αυτά θα πρέπει να ε, ολοκληρώσουμε. σε σχέση με τους στρατηγικούς μας στόχους ως Ευρώπη, αλλά να ωφελήσουμε και τους Αφρικανούς και να επικεντρώσουμε τις προσπαθειές μας στους νέους, να δώσουμε ευκαιρίες στις νέες γενιές. Αυτό είναι το πιο σωστό. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και για τα δημογραφικά προβλήματα της Αφρικής. Για τα οικονομικά προβλήματα. Να καλύψουμε τους Αφρικανούς είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση κορυφής που θα γίνει σε μόλις λίγους μήνες. Θα προεδρεύσει ο κύριος Τούσκ, αλλά θα συμπροεδρεύσει και ο Αφρικανός ομολογός. Οπότε και εμείς θα διευκολύνουμε, θα προπαρασκευάσουμε τη συνάντηση κορυφής. θεματολόγιο που θα περιέχει καινοτομίε όπως τα ψηφιακά, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Να δώσουμε ευκαιρίε στη νέα γενιά, αλλά να γίνουν και υπόλογε οι κυβερνήσει, να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια. Τώρα, για Κονγκό και Νιγηρία... Είπαμε, όλα τα μέσα να χρηματοδοτούνται. Ρίξτε μια ματιά τι γίνεται όσον αφορά τα στοιχεία. Κοιτάξτε τι γίνεται με τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, κρατών μελών. Ε, υπάρχει αύξηση. Απλώς έχει αυξηθεί και η ζήτηση. Πολύ περισσότερο από την προσφορά. Ιδίως για την ε, Νιγηρία σε σχέση με την Μπόκο Χάραμ και συναφείς συμμορίες. Άρα θα πρέπει για αυτά τα προβλήματα να βοηθάει κανείς τον κόσμο που πλήσεται. Και σε πολλές περιπτώσεις ε, ακόμα πιο δύσκολο να, να παρέμβει σε τέτοιες κρίσεις ε, παρά το να βρει τα χρήματα είναι θέμα της ανθρωπιστικής ασφάλειας εν προκειμένου. Α, τώρα απαντώντας κάλυψα ε, εν μέρη τον κύριο Νόζερο όσον αφορά την ασφάλεια σχέση με Αφρική. Επίσης υπήρχε και μια ερώτηση σε σχέση με την περίοδο μετά την Κοτονού πλησιάζει η δεκαετία ε, του 2020. Έχουμε κάποιες προτάσεις για τη σχετική εντολή. Έχει συζητηθεί μια σχετική ρύθμιση από το Συμβούλιο και μπορώ να σας πω τώρα δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει 100% αλλά εμείς είμαστε ε, τώρα ε, είμαστε ταγμένοι σε αυτή την προσπάθεια να βρούμε μια συνένεση και έτσι να υπάρξει ένα τέτοιο θεματολόγιο για τη σχέση με την Αφρική. Αυτό είναι προτεραιότητα και συνεχίζουμε πάντως να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας από Καραϊβική και Ειρηνικό αναζητούμε τρόπους λοιπόν ούτως ώστε να εμπλέξουμε και άλλους περιφερειακούς εταίρους στην περιοχή του Ειρηνικού και στην Καραϊβική για συγκεκριμένα συμφέροντα να υπάρξει συγκεκριμένη βοήθεια για αυτό το θεματολόγιο σε σχέση με αυτές τις ε, ομάδες χωρών και ελπίζουμε αυτά να τα συζητήσουμε και να τα συμφωνήσουμε πριν εκπνεύσει η ισχύουσα ρύθμιση να σημειώσουμε πρόοδο ελπίζουμε να μην πάει χαμένη η πολύτιμη κτήθησα εμπειρία και όλα τα μέσα πολιτικής που έχουν ε, θεσπιστεί και χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Α, για την Ιταλία. Και το μεταναστευτικό. Ε, ε, βέβαια και είναι σοβαρή η κατάσταση. Τα συζητήσαμε και στην ΑΦΕΤ χθες. Είναι αυτό το θέμα της ε, διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου. είναι ένα από τα βασικά θέματα ασφάλειας. Αυτό θα συζητείτε τους αμέσως επόμενους μήνες από την Προεδρία μας και σε περισσότερα από ένα συμβούλια γιατί υπάρχουν θέματα εδώ εξωτερικής ασφάλειας, εξωτερικών σχέσεων αλλά και εσωτερικής ασφάλειας. Είναι και θέμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Ε, βέβαια, και θα πρέπει να δούμε τι απαιτείται να γίνει άμεσα και θα πρέπει στα σοβαρά να λάβουμε υπόψη το Ιταλικό αίτημα προς αλληλεγγύη από πλευράς κρατών μελών. Επίσης να αναζητήσουμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε μακρόπνο και στρατηγικά το πρόβλημα. καταπολεμώντας τις συμμορίες τους εγκληματίες που εποφελούνται και παράνομα διακινούν τον κόσμο εκεί. Να γίνει καταγραφή των μετακινουμένων, να βρούμε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για το θέμα. Και θα πρέπει στα πλαίσια εξωτερικής πολιτικής να δούμε τις Αιτίε τη μεταναστευση. Ε, και εδώ βέβαια είναι θέμα ανθεκτικότητα και αντοχής. Να βοηθήσουμε δηλαδή ουσιαστικά, ούτω ώστε να αυξηθούν οι ικανότητες και οι δυνατότητες των χωρών διαμετακόμισης αλλά και προέλευσης των μεταναστών για τα σύνορά τους, γενικά για την κατάσταση της μετανάστευσης. Επομένως, είναι πάρα πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Υπήρξε προτεραιότητα το μεταστευτικό και στην Μαλτέζικη Προεδρία. Γίνανε βήματα πρόοδο, αλλά βέβαια και δεν μπόρεσαν να λύσουν 100% το πρόβλημα. Και όχι επειδή δεν προσπάθησε η Μαλτέζικη Προεδρία, αλλά διότι η κατάσταση είναι τόσο περίπλοκη. Εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας, τόσο ώστε να προωθηθεί το ζήτημα. Και ελπίζουμε να τελειώσει η δική μας Προεδρία, να είναι τα πράγματα καλύτερα. Τότε είναι και εποχιακό θέμα μετανάστευση στην Κεντρική Μεσόγειο, οπότε έχουμε τότε και τα Χριστούγεννα αλλά θα είναι καλύτερα τα πράγματα γιατί ελπίζουμε να έχουμε πλησιάσει σε μεγαλύτερη συνένεση για τα θέματα ευθύνης και ελληνική μεταξύ κρατών μελών. Ε, βέβαια και θέλουμε να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί διαμεσολαβητές και θα αφιερώσουμε κάθε ικμάδα δύναμης προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε τον αξιότιμο κύριο Υπουργό γιατί προσπάθησε να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα τα οποία ήταν απαραίτητα για την ενημέρωση της Επιτροπής μας. Είναι έξι μήνες που διαμεσουλαβούν μέχρι τα Χριστούγεννα και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ και που ήρθατε να μας δείτε και που τηρήσατε το χρόνο. Ένα-δύο λεπτά διακοπή για να έχουμε τα καρτελάκια με τα ονόματα των επόμενων ομιλητών. Okay, Συνάδελφοι, προχωρούμε στο σημείο 9 της ε, ημερήσιας διάταξης, ενδιάμεση επανεξέταση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε, έχουμε περάσει τα μισά της κοινοβουλευτικής θητείας, τρία χρόνια από την πρώτη μέρα που τα είπαμε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Άρα, και τα εργαλεία μας είναι στα μισά του δρόμου, στα μισά της διαδρομής και είναι ευκαιρία η Επιτροπή μας να επανεξετάσει αυτά τα εργαλεία και να δει κατά πόσο πρέπει να γίνουν αλλαγές. Για να το αποφασίσουμε πρέπει να αξιολογήσουμε το πώς δουλεύουν τα πράγματα, πώς λειτουργούν και θα ακούσουμε σήμερα τις αξιολογήσεις που έκαναν για χάρη της Επιτροπής μας οι εμπειρογνώμονες. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες θα μιλήσουμε για το ΜΑΣ και το ΕΤΑ. Το Ζόμπο Σούτ έχουμε μαζί μας, το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας και το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Έχουν κάνει ε, πολλές μελέτες στο παρελθόν. Η κυρία Κάρολιν Τουνίσεν και ο κύριος Χαβιέ Περέιρα θα μας μιλήσουν για το ΕΤΑ που είναι σύμβουλοι με πολύ μεγάλη εμπειρία, χρόνια στη συμβουλευτική σε θέματα ανάπτυξης και αναπτυξιακά γενικότερα. Να ξεκινήσουμε με το ΕΤΑ λοιπόν. Οκτώ λεπτά έχετε και οι δυο σας, Καρολίν και Χαβιέ. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου ομιλήτρια. Τώρα με ακούτε. Ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θα παρουσιάσω τα βασικά συμπεράσματα σε οκτώ ε, λεπτά του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου Υπαριθμών 11 θα ήθελα να σας ε, δώσω το πλαίσιο. Είναι ένα από τα εννέα εξωτερικά εργαλεία, εργαλεία εξωτερικής χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 30,5 δις ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι ένας από τους μεγαλύτερους φακέλους ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Δίδεται εντός πολιτικού πλαισίου που είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού και γι' αυτό έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρέπει να υπάρχει εταιρική σχέση και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών που δικαιούνται αυτή την στήριξη και αυτή τη βοήθεια. Και γι' αυτό επειδή είναι εταιρική σχέση οι ενδιαφερόμενες χώρες πραγματικά οικειοποιούνται το πρόγραμμα, και το προσυπογράφουν και συμφωνούν με αυτό. Ε, έχουμε την ομάδα υψηλού επίπεδου για τη στρατηγική πολιτική και για το διάλογο που προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες. Τρίτο χαρακτηριστικό, η γεωγραφική σκοπιά του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογή σε πάρα πολλές χώρες, 25 εξωχώρες, εξόχως απόκορα, κέντρες Αφρική, Καραϊδική, Ειρηνικός και έχουμε σε επίπεδο εθνικό, επίπεδο περιφερειακό και επίπεδο ενδοακέ είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα σε όλες αυτές τις χώρες. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης έχει το ΕΤΑ το δικό του κανόνα για την εφαρμογή του. Ε, έχουμε πολύ ευρεία σειρά εργαλείων και πολλές, πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και λεπτομέρειες εφαρμογής όλων αυτών, ε, διότι μιλούμε για απίστευτα πολλά χρήματα και για πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις χώρες όπου ενεργοποιείται. Υπάρχει νομικό πλαίσιο μακροπρόθεσμο 5 με 7 χρόνια, η τελευταία περίοδος είναι 7 ετών και άρα είναι ένα πολύ προβλέψιμο εργαλείο με την συνεχή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα. Τι κάνει. Στηρίζει τη μείωση της φτώχειας, στηρίζει την αηφόρο και ισότιμη ανάπτυξη, δίκαιη για όλους προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες και συμπληρώνει και άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά για να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικές προκλήσεις της οικονομίας. Μιλούμε δηλαδή για ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λύνοντας τα διαρθρωτικά προβλήματα και εκεί όπου χρειάζεται να αντιμετωπιστούν επίγουσες ανάγκες, τότε άλλα εργαλεία εξωτερικής χρηματοδότησης ενεργοποιούνται και όχι αυτό. Αυτό που το καθιστά μοναδικό, το έτα, είναι ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συγκεντρώνονται και ε, του δίνουν τη δική του προσωπική χρειά. Έρχομαι τώρα στα ευρήματα και στα βασικά συμπεράσματα της αναθεώρησης, η οποία διαιρείται σε τέσσερα κεφάλαια. Τα δύο πρώτα έχουν να κάνουν με τις επιδόσεις του εργαλείου, το πώς λειτουργήσε και τα δύο τελευταία κεφάλαια έχουν να κάνουν με τη διάρθρωση, τη δομή, την διοργάνωση, την αναδιοργάνωση και τα εργαλεία που αξιοποιεί το ΕΤΑ. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται η αναθεώρηση στα μέσα του 2016 και ολοκληρώθηκε στα 2017 στις αρχές, είναι ότι μόλις τότε έχει αρχίσει να ε, εφαρμόζεται και γι' αυτό λίγα μπορούμε να πούμε για την αποτελεσματικότητά του. Άρα η αξιολόγηση σε κατά βάση στηρίζεται στο προηγούμενο, στο δέκατο έτα και όχι στο ενδέκατο που ισχύει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε και εξετάζουμε κατά πόσο η δομή και η διάρθρωση ταιριάζει για να είναι αποτελεσματική η βοήθεια που δίδεται στους δικαιούχους. Εδώ η ερώτηση που τίθεται είναι πώς το EDF το ε, ΕΤΑ 11 ταιριάζει και αλληλεπιδρά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και πόσο ταιριάζει με το πολιτικό και αναπτυξιακό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση είναι καταφατική, παρόλο που ο κόσμος αλλάζει συνεχώς και παρόλο που έχουν προκύψει νέες προτεραιότητες, είναι ένα εργαλείο που μας έχει βοηθήσει, έχει χρησιμεύσει και έχει λειτουργήσει πολύ καλά. έχει ε, ε, αντιμετωπίσει τις βασικές ε, προτεραιότητες, έχει συμβάλει στα αναπτυξιακά αποτελέσματα, έχει εφαρμόσει τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και άλλες γενικότερες αρχές με μικρότερη και μεγαλύτερη επιτυχία. Έχει αποτελέσει ένα καλό σημείο εισόδου για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών όπως είναι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής και την ενσωμάτωση τέτοιων διαστάσεων σε όλους τους κλάδους και τους τομείς και τα πεδία που επιλέγεται να χρηματοδοτήσει και να στηριχθούν. Και τέλος, μας ταιριάζει αυτό το εργαλείο στους στόχους για την αηφόρο ανάπτυξη και για το νέο διεθνές θεματολόγιο που περιλαμβάνει θέματα όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια και πρέπει να βασιστεί σε ένα καταπίστευμα για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς τους, του και η χρήση του καταπιστεύματος του Trust Fund έχει επιπτώσεις ε, για τις ε, θεμελιακές του αρχές και την αποτελεσματικότητα. Δεύτερη ερώτηση. Πώς θα πήγε το εργαλείο αυτό με την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών, γιατί σας μίλησα για την εταιρική σχέση, για τη συνεργασία και για τη διοκτησία του εργαλείου από πλευράς ε, τρίτης χώρας που δέχεται αυτή τη βοήθεια. Είναι εργαλείο σε βάθος χρόνου με ορίζοντα 7 ετίας και άρα λειτουργεί ως άγκυρα από την οποία αγκιστρώνεται το κράτος που είναι δικαιούχος. Είναι μια απάντηση ε, σταθερή στις αναπτυξιακές προκλήσεις με προβλεψιμότητα. Αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι καλό για τους γνωστούς λόγους, αλλά γιατί είναι και κακό γιατί δυσκολεύεται το εργαλείο αυτό να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες. Κάποιες δράσεις είχαν προγραμματιστεί πολύ καιρό πριν και όταν εφαρμόζονται τελικά ίσως είναι άσχετες και δεν ταιριάζουν τόσο με τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Ένα από τα βασικά ευρήματα της αναθεώρησης είναι το εξής. Οι αρχές εταιρικής σχέσης δεν έχουν προωθηθεί έτσι περαιτέρω παρόλο που αυτό ήταν ρητή, ρητός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λιγότερη και μικρότερη εταιρική σχέση και λιγότερη και μικρότερη ιδιοκτησία, διότι για τις επιλογές του προγράμματος οι αποφάσεις ελήφθηκαν στις Βρυξέλλες και αυτό ε, ε, εντάθηκε λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης στους διαφόρους τομείς. Ε, είναι καλό να υπάρξουν απλουστευμένες διαδικασίες, να προσφύγουμε στο καταπίστευμα, να υπάρχουν μίξες. Όλα αυτά θεώρησαμε ότι είναι καλό, αλλά από την άλλη υπάρχουν λιγότερες εταιρικέ σχέσεις με τις χώρες που είναι εταίροι μας. Και γι' αυτό ενδεχομένως ε, προέκυψαν διάφορα προβλήματα με τη δομή των εθνικών γραφείων που εξουσιοδοτούν και δίνουν το πράσινο φως, είναι οι συνομιλητές μας στις χώρες δικαιούχους και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαβρυνθεί η εταιρική σχέση. Δηλαδή η εταιρική σχέση γίνεται με την κυβέρνηση και έστω με ε, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τις ΜΚΟ κτλ. Αλλά όχι σε αρκετό βάθος. Και γι' αυτό ε, χρειαζόμαστε να εμπλακούν και π.χ. πολιτικά κόμματα ή θρησκευτικοί ηγέτες, άλλα τμήματα και εκπρόσωποι της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στις κατατόπους χώρες δικαιούχους. Ας δούμε λοιπόν ε, πώς ταιριάζει με το σκοπό. Αν ταιριάζει με, για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με το συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει διάφορα βήματα για να διασφαλίσει ότι η αυξημένη συμπληρωματικότητα και ο συντονισμό μεταξύ των ε, διαφόρων έργων, προγραμμάτων και εργαλείων και η πρόκληση είναι ε, το γεγονός ότι διαχειριζόμαστε κεντρικά τις γραμμές του προϋπολογισμού. Άρα είναι αδύναμες οι συνέργειες των δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο εντός ΑΚΕ. Άρα εδώ είναι ένα πεδίο που μπορεί να σημειωθεί και πρέπει να σημειωθεί πρόοδος. Στην πρώτη διαφάνεια σας μίλησα για τις διάφορες πτυχές και τα διάφορα χαρακτηριστικά του εργαλείου που θα έπρεπε να το μεταμορφώσουν σε κάτι το καταπληκτικό, να μας βοηθά να έχουμε ενεργητική δράση υπέρ της ανάπτυξης, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει αξιοποιήσει πλήρως και δεν το έχει εκμεταλλευτεί πλήρω, δεν έχει εκμεταλλευτεί όλε τι δυνατότητε αυτού του καταπληκτικού εργαλείου. Την η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια προσέγγιση του στυλ ένα νούμερο να ταιριάζει σε όλου, ένα ε, πλαίσιο να ταιριάζει σε όλου, χωρί να λαμβάνει υπόψη τι εκάστοτε ιδιαιτερότητε των τρίτων χωρών, των χωρών εταίρων και πολύ συχνά αξιοποιείται για να γίνεται πολιτικός διάλογος και διάλογος για τη χάραξη πολιτικής. Τέλος, και ελπίζω να μην έχω ξεπεράσει το χρόνο που μου έχετε δώσει κυρία Πρόεδρε, τίθεται ένα τελευταίο ερώτημα, ποια εργαλεία έχει στη διάθεσή του το συγκεκριμένο εργαλείο, το ΕΤΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, για να πετύχει τους στόχους. Πρώτο συμπέρασμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις προσπάθειες να αυξήσει και να ενισχύσει και να βελτιώσει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ε, παραμένουν οι ελλείψεις ό,τι έχει να κάνει με τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση των πόρων, τα αμετρήσμα μετρήσιμα αποτελέσματα με βάση δικτών, ουσιαστικά μετρά το επίπεδο συμμόρφωσης, άρα η παρακολούθηση ή η αξιολόγηση περιορίζει τη δυνατότητα του εργαλείου να παρουσιάζει αναφορά του πόσο αποτελεσματικό είναι το ίδιο και μειώνεται και η λογοθεσία στους πολίτες Περιορίζεται δηλαδή η λογοδεσία προς όλους και οι δυνατότητες να αντλούνται διδάγματα για τον μελλοντικό σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων. Αυτά δηλαδή είναι λίγο προβληματικά. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολλές προσπάθειες να πλουστεύσει τις διεργασίες, τις διαδικασίες και να ενοποιήσει όλα αυτά τα εργαλεία εξωτερικής χρηματοδότησης έτσι ώστε να υπόκειται στους ίδιους κανόνες. Είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια. Είδαμε κάποια θετικά στοιχεία, δεν είδαμε το άμεσο αποτέλεσμα ακόμα. Περιμένουμε ότι μειώνεται ο διοικητικός φόρτος, έχουμε καλύτερη οικονομική επίδοση, όμως αυτές οι διαδικασίες απλούστευσης πέρα από τα ε, ε, ε, ευεργετήματα έχουν και αρνητικά, γιατί είναι πρόβλημα το, η πρόσβαση του CSO σε χρηματοδότηση. Είναι περισσότερο, δηλαδή, γίνεται περισσότερο διαχείριση και όχι συνεργασία για ζητήματα φλέγοντα επί τόπου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, η Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις θα έχουμε στην επόμενη παρουσίαση. Ο κύριος Μποσιού να πάρει το λόγο για το ΜΑΣ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία είναι όπως ε, το Ταμείο Ανάπτυξης, γι' αυτό τα έχουμε σε κοινή συζήτηση αφορά και άλλες χώρες ε, ε, ε, στην Ασία και στην Λατινική Αμερική και έχει και διμερεί προγράμματα για τις χώρες αυτές, αλλά έχει και τρία θεματικά προγράμματα που κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με την αξιολόγηση θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Είναι το πρόγραμμα για την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης, ένα πρόγραμμα για τα δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις, πριν από το θεματολόγιο του 2030 και σύμφωνα με την αξιολόγηση αποτελεί ένα πρόδρομο όλων των καινοτομιών και ένα τρίτο στοιχείο ε, αφορά την Αφρική ε, με δράση στην Ευρώπη και στην Αφρική. Παρόμοιες δράσεις όπως και των φίλων μας από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία αποδείχθηκε αποτελεσματικό όσον αφορά τη συνεργασία με περισσότερο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερο σχεδιασμό και για να επιτύχουμε την, το θεματολόγιο της αλλαγής του 2011 και τη διαφοροποίηση μας βοήθησε πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα μέλη του κόσμου όπως η ε, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Βραζιλία, διαφορετικές χώρες ε, με διαφορετικά στοιχεία της, ε, του θεματολογίου της αλλαγής, απελευθερώνοντας σπόρους για τις πιο ευάλωτες φτωχές χώρες. Με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα λοιπόν αυτό το μέσο κατάφερε να λάβει υπόψη του νέες ε, ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη. Δεν ήταν εύκολο για το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας να λάβει υπόψη και άλλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και για το Ταμείο Αναπτυξιακής Βοήθειας. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραδείγματος χάρη, είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε τέτοια μέσα για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου ή και για την ε, προώθηση των ε, δημοσίων αγαθών. Μέσω των διμερών προγραμμάτων δεν είναι εύκολο να προωθήσουμε την κλιμα... μέτρα για την κλιματική αλλαγή ή άλλες παγκόσμιες προτεραιότητες. Όσον αφορά λοιπόν την αποτελεσματικότητα, τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντοτε άριστα. Είναι ένα σύνθετο έργο με πολλές συνιστώσεις και γι' αυτό δεν ήταν εύκολες οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα. Συνυπήρχαν οι διάφορες συνιστώσεις και η συνέργεια μεταξύ αυτών αποτελούσε πρόκληση. Όσον αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, υπήρχε κάποια πρόοδος για τον κοινό προγραμματισμό, αλλά ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η ερώτηση είναι τι κάνουμε με τέτοιου είδους μέσα, τι προσφέρουν στην Ευρώπη. Για το Ταμείο Αναπτυξιακής Συνεργασίας είπατε ότι υπάρχουν πολλά κονδύλια. Τώρα όσον αφορά το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας δεν ήταν τα χρήματα ο κύριος παράγων όθησης. Υπήρχαν όμως πάρα πολλές χώρες η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν τόσο ο όγκος των κονδυλίων, αλλά το ότι θεωρείται περισσότερο ουδέτερος ε, υπερεθνικός φορέας με, μια, με ένα θεματολόγιο περισσότερο ουδέτερο και αυτό είναι συμπληρωματικό ως προς το έργο των κρατών μελών. Επίσης, Άλλο ερώτημα ήταν αν τα χρήματα τα οποία διατίθεται μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μόχλευση ώστε να κινητοποιήσουν κονδύλια και από τον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ η απάντηση είναι θετική. Δηλαδή είχε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα περισσότερο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και συνεργασία. Ήταν πολύτιμο αυτό το μέσο για την ε, μείωση της φτώχειας σε ευάλωτες χώρες σε πολλά σημεία του κόσμου. Πολλές από τις ε, χώρες αυτές σιγά σιγά ε, γίνονται χώρες μεσαίων εισοδημάτων ή και στο επάνω στρώμα των μεσαίων εισοδημάτων, οπότε βγαίνουν σιγά σιγά από την αναπτυξιακή βοήθεια, άρα αυτό το μέσο δεν ήταν σχεδιασμένο πια για αυτές, άρα δεν είναι πια ελκυστικό μέσο για τις χώρες αυτές. Οπότε δημιουργείται ένα κενό στη δέσμη των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και αυτό σιγά σιγά θα ισχύσει και για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο όσο οι χώρες βγαίνουν από την αναπτυξιακή βοήθεια. Η αξιολόγηση λοιπόν το 2017 εντοπίζει ένα κενό στην κάλυψη χωρών. Δηλαδή οι χώρες αυτές δεν χρειάζονται αναπτυξιακή βοήθεια και δεν λαμβάνουν και πλέον αναπτυξιακή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της πολιτικής της. Πώς να έχουμε όμως ένα χαρτοφυλάκιο συνεργασίας με βάση το βαθμό ανάπτυξής τους και με βάση τις ε, δυνατότητε των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το καλύψει το μέσο ανεπτυξιακής συνεργασία αυτή τη στιγμή και υπάρχει ακόμη αυτό το κενό. Όπω και για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, παρόλε τι προσπάθειες γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και τι τοπικέ κοινότητε. Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για, την, για το θεματολόγιο του 2030 βάσει των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς να έχουμε αυτό το άνοιγμα προς την κοινωνία των πολιτών και την πολυμερή συνεργασία. Και κλείνοντα, ένα σημαντικό σημείο ότι το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία μπορεί να παραμείνει ενδιαφέρον μέσο, τουλάχιστον λόγω των γεωγραφικών συνιστοσών του, να παραμείνει για αυτές τις φτωχέ ευάλωτε χώρε. Δεν ξέρω κατά πόσο τα δύο μέσα στο μέλλον θα συζητήσετε να, να ε, συγχωνευτούν. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για όλες αυτές τις χώρες. Μιλάμε για ερωτήματα που θα πρέπει να τεθούν στο μέλλον για να αναβαθμιστούν τα μέσα που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε στο μέλλον να συνεργαστούμε με τις χώρες που είναι ε, μέσων εισοδημάτων ή ε, ε, στο ανώτερο επίπεδο των μέσων εισοδημάτων. Αυτά τα ερωτήματα θέτω προς συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κρατήσατε και τον χρόνο σας. Θα δώσουμε το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε τώρα το λόγο. Όχι, ας ακούσουμε ερωτήσεις των κρατών μελών. Ας, ε, τον, θα ε, ακούσουμε τις ε, ερωτήσεις των κυρίων βουλευτών. Και δίνω το λόγο στην Μαρία Χόιμπουρ καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε για τις αξιολογήσεις. Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και για τις προτεραιότητες μέσω του καταπιστευματικού ταμείου. Η ενδιάμεση αξιολόγηση έχει, μιλάει για ένα ε, αποθεματικό και καταλήγει μετά την ανάλυση ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με την διαφάνεια, με την ανάληψη και το κατά πόσο ενστερνίζονται οι χώρες της Αφρικής αυτά τα προγράμματα. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πώς θα διασφαλίσουν ότι θα ακολουθήσουμε την αρχή ε, της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας. Και τα χρήματα και οι πόροι για τις ε, τωρινές ε, προτεραιότητες πιστεύετε ότι καλύπτουν τις ανάγκες. Έχω θέσει και γραπτός μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αξιολόγηση. Και στην απάντηση Η Επιτροπή δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη στην αξιολόγηση και θα παραμείνει σε επαφή με τους αξιολογητές για να κατανοήσει καλύτερα τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να μου πείτε πού υπήρξε κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν είχε κατανοήσει σαφώς η Επιτροπή τα αποτελέσματα. Θα ήταν ενδιαφέρον να καταλάβουμε τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Στα συμπεράσματα που μας παρουσιάσετε για το μας, ιδίως εν τέλει, πρόγειψε ότι είναι πάγιο θέμα ζήτηση στην Επιτροπή μας. Δηλαδή, το πώς θα συνεργαστούμε με χώρες μέσου εισοδήματος ή τέλο πάντων μέσου προς τα επάνω. Και πάγε γίνεται η συζήτηση για το τι μέσον υπάρχει για την μέτρηση του εισοδήματος. Τι είναι, είναι κάποιος ε, στατιστικός δείκτης ε, κάποιος μέσος όρος, όμως πολλές φορές οι μέση όροι αποκρύπτουν κάποιες σημαντικές ανισότητες. Μπορεί να είναι μεταξύ περιφερειών αυτές οι ανισότητες, μεταξύ ε, μειονοτήτων, μεταξύ ηλικιακών κατηγοριών, μεταξύ ε, εισοδηματικών κατηγοριών, κάθε είδους. Ή για διάφορους λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει συμφέρον να συνεργαστεί δέσμευσε να συνεργαστεί με κάποιες χώρες που επί τη βάση αυτών των δικτών βρίσκονται στα όρια ή εκτός ορίων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά διευρύνουμε το θέμα και αντιμετωπίζουμε, θα έπρεπε να τέλο πάντων την εσωτερική περιπλοκή της χώρας ε, ούτω ώστε να έχουμε κάποιο είδου ε, πρωτοβουλίες δικές μας να κάτσουμε δηλαδή και φάντας να δούμε το πώς θα συνεργαστούμε με αυτά τα μέσα πολιτικής. Πρόεδρος. Έχω και εγώ μια διερώτηση. Αν έλεγε κανείς στην Επιτροπή, αλλάξτε κάποια πραγματάκια. Είναι τεράστιο αυτό το πρόγραμμα, είναι πάρα πολλά έργα, projects υπάρχουν. Υπάρχει συνένεση για τα SDG. και για το τι χρήζει χρηματοδότησης. Έχουμε διάφορα ταμεία, διάφορους πόρους, έχουμε τα διαρκτικά ταμεία, έχουμε ε, ε, ταμείο για, και πόντους για χώρες που ας πούμε, χρειάζονται βοήθεια όσον αφορά το νερό ή τη βιομηχανία απασχόληση. Τα έχουμε αυτά και στο ιστορικό τη Ένωση. Έχετε να κάνετε κάποια σύσταση. Μα γι' αυτό έγινε αυτή η αξιολόγηση. Για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Και για το μας και για τα άλλα μέσα. Τι μεταβλητές διαβούν τη σχέση δωρητή και αποδέκτη. Συγκεκριμένα. Τι, τι, τι ισχύει, γιατί στις συνεδριάσεις σαν τη δική μας έχουμε ένα σωρό όρους ξύλινης γλώσσας. και εξειδικευμένης ορολογίας. Λοιπόν, για πέστε μας συγκεκριμένα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχετε το λόγο. Α, μήπω να ζητήσουμε να μας μιλήσει πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν είναι εσείς. Πες μας τι θα κάνετε εσείς με την αξιολόγηση και μετά να μα πούνε οι ειδικοί. Και έτσι θα τα σκεφτούν κιόλας, θα έχουν χρόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτές οι αξιολογήσεις βοηθούν για την προπαρασκευή της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης και αναθεώρησης Είναι εξωτερική αξιολόγηση ανεξάρτητη. Ολοκληρώθηκε τώρα. Δημοσιοποιείται. Οπότε τώρα έχουμε πολλά να μας απασχολήσουν, να προβληματιστούμε. Και μια της προκλήσεις είναι ότι όταν είναι θέμα ταμείων άπτυξης ή μέσω συνεργασίας τότε θα πρέπει να μπορεί κανείς να δει αν είναι τα πιο δόκιμα για την επιτεύξη των σκοπών αυτά τα μέσα στο συγκεκριμένο πολιτικό κύκλο. Νομίζω τώρα είναι ξεκάθαρο το ότι απόψεις διαμορφώθηκαν. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Δεν έχουμε πάντα δεδομένα και στοιχεία. Το έχουμε πάντα τα μέσα υποστήριξη αυτών των αξιολογήσεων. Τέλος πάντων, μια επιλογή που κάναμε εμείς. Είναι στον αιτήσιο προπολογισμό να καλύπτουμε αυτά τα μέσα μας και τα. Έχουμε διάφορα μέσα πέραν αυτών στον προπολογισμό. Αλλά για το EDF υπάρχει διαφορετική νομική διαδικασία. Θέλουμε πάντως να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτές τις ε, προσπάθειες και αξιολογήσεις. Να συγκρίνουμε δηλαδή τα διάφορα μέσα και να δούμε τι αποκομίζουμε. Παρά τις διαφορές τους. Ε, τι θα πρέπει να κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες. Θα πρέπει να κάνουμε μια έκθεση λογικής συνοχής. Συνθετική εργασία. Για τις επιμέρους αξιολογήσεις. Να, κι άλλο υλικό πέραν των αξιολογήσεων. Έχετε πολλά να μελετήσετε, αλλά σας καλώ να διαβάσετε και αυτή την έκθεση συνεκτικότητας. Δηλαδή, τι συνέργειες υπάρχουν μεταξύ των επιμέρους μέσων, τι Άλλα προβλήματα υπάρχουν τώρα. Και αυτό είναι πολύτιμο όταν κανείς έρθει η ώρα να παρέμβει σε συγκεκριμένη χώρα και περιοχή φέρει. Είπαμε ότι είχαμε αυτού του είδους την ε, διαδικασία διαβούλευσης του τριμήνου Θα πρέπει δηλαδή να δούμε τι πρόκειψε αυτή τη διαβούλευση. Τέλος του Μαρτίου είχαμε εκείνο το τεχνικό εργαστήρι και εσείς είχατε συμμετάσχει και τα κρατημέλη. Διάλογος και διαβούλευση. Πολύ σημαντικά αυτά για να μπορέσουμε να προβληματιστούμε. Και το επόμενο βήμα εμείς η εξωτερική υπηρεσία είναι να έχουμε κάποια υπηρεσιακά κείμενα. Λαμβάνω πως εξολογίζεις αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να τοποθετηθούμε επ' αυτών. Staff Working Documents λέγονται. Και κατόπιν έχουμε τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση για τη σχετική έκθεση του Δεκεμβρίου. Να τα επόμενα βήματα και έτσι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτήν την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση. Α, το Δεκέμβριο επομένω θα έχουμε νέα. Ναι, ναι, τελευταία φορά κάνατε κάτι αλλαγές. Ωραία. Και τώρα ο λόγος τους εμπειρογνώμονες. Thank you very much. I'll launch into the, the first. Uh, I think I'll keep <laughs> your global question uh, for the end. Uh, in terms of the trust fund... Όσον αφορά τα καταπιστεύματα, συμφωνήσαμε Ήδη το είχαμε συζητήσει όσον αφορά τη βασική διαφορά μεταξύ των απόψεων της Κομισιόν και των συμβούλων. Από πλευράς νομικής κοιτάξαμε αυτά τα καταπιστεύματα. Και ήταν σαφές ότι δεν υπήρχαν τίποτα ειδικοί κανόνες όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για αυτά τα καταπιστεύματα. Και από το EDF δόθηκαν κάποιοι πόροι σε κάποιο καταπίστευμα. Παρ' όλα αυτά, από πλευράς Επιτροπής, τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Και επομένως οι συνεργαζόμενοι θα ήθελαν να συνεχθεί μαζί του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Και κάναμε μία αξιολόγηση επιδόσεων. Όχι του καταπιστεύματος, αλλά του Ταμείου ανάπτυξη. Οπότε αυτό το οποίο προτείνουμε στην εκκλησία μας είναι να γίνει ανεξάρτητη αξιολόγηση των καταπιστευμάτων. Οπότε να δούμε όλα τα θέματα από πλευράς νομικού πλαισίου. Οπότε είδαμε τα διάφορα ζητήματα της εταιρική σχέσης, της βιωσιμότητας, της αποτελεσματικότητας. Μην ξεχνάτε ότι η αξιολόγηση μας και το καλοκαίρι του 16 και είχαμε και την διάμεση έκθεση μετά το Φεβρουάριο του 2017. Οπότε είχαμε ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Και είχαμε και τις δημοσίευσεις για τα καταπιστεύματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε στην τελευταία έκθεση αυτά διορθώθηκαν. Αυτά, αυτά. Τώρα, για το τι θα κάνουμε για τις χώρες μέσα εισοδήματος. Δεν ζητήθηκε να τα να αποφανθούμε γι' αυτό. Άμα κοιτάξετε τις συστάσεις μας θα καταλάβετε. Τι πιστεύουμε. Είναι σημαντικό το ότι εάν θέλει κανείς να συνεχίσει το Ταμείο Ανάπτυξης να αποτελέσει μέσω συνεργασίας, ε, τότε θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια ανανέωσης, ανακαίνησης της σχέσης με εκείνες τις χώρες και πιο δημοκρατική δημοκρατικότητα του να διέπει την συνεργασία. Να είναι διάλογος όχι μόνο με τις κυβερνήσεις, αλλά να είναι διάλογος με περισσότερη συμμετοχή διαφορετικών στρωμάτων της κοινωνίας. Και έτσι να κρίνεται προς τα που θα πάει η ανάπτυξη. Δεν υπάρχει καμία έτοιμη εύκολη λύση. Πάντω αυτό που ζητήσατε για τι χώρε μεσαίου εισοδήματο δεν το... Δεν μας είπατε το αντιπαντήσω. Ευχαριστώ. Να σα πω ότι και το ΜΑΣ και όλα τα εργαλεία έχουν συμβάλει σε αυτό που λέτε. Τι σημαίνει όμως όλο αυτό είναι ένα σύστημα, ένα σχέδιο που προκύπτει από όλες τις αξιολογήσεις. Δηλαδή, ο όρος ευελιξία επανέρχεται ξανά και ξανά. Θέλουμε καταπιστεύματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να δώσει πολιτική απάντηση σε διάφορες προτεραιότητες και πρέπει να κινητοποιήσει διάφορα κονδύλια και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Έχουμε τα δύο εργαλεία στην αναπτυξιακή συνεργασία, το core και το partner και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και άλλα συμφέροντα και άλλα ενδιαφέροντα πρέπει να ικανοποιηθούν. Έχουμε τα αμοιβαία συμφέροντα όπου δεν έχουμε πλέον δωρητές και παραλήπτες βοήθειες, αλλά έχουμε θεματολόγιο εταίρων και έχουμε και συμφέρον ε, ε, εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βρίσκουμε μέσα στο μας το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας ότι συμφιλιώνουμε διάφορες πολιτικές επιδιώξεις την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ασφάλεια, την επίλυση της προσφυγικής κρίσης και του καθεξής στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά έχουμε και αμοιβαία συμφέροντα. Αυτό είναι διαφορετικό είδος συνεργασίας και μετά έχουμε και εσωτερικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για να συμφιλειωθούν όλα αυτά, να ταιριάζουν άλληλο, διαρθρώνονται και να γίνεται σωστή συναρμογή, επιλέγεται η μορφή των καταπιστευμάτων, trust fund. Και πρέπει να βρεθούν τα κατάλληλα σημεία ισορροπίας και τώρα και στο μέλλον. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα του κυρίου Γκερέρο. Ήταν δύσκολο αυτό που αναφέρεται για το, για ΜΑΣ, γιατί το θεματολόγιο για την αλλαγή θέσπισε την αρχή της διαφοροποίησης και έγινε μακρά συζήτηση εδώ για όλα αυτά. Κάποια στιγμή η βοήθεια δεν είναι λύση και εργαλείο για να δουλέψουμε με αυτές τις χώρες και σαφέστατα επιλέγονται δείκτες και μπορεί κανείς να συζητά ατέρμονα για τους δείκτες, όμως η έκθεση του μας λέει ότι ίσως η αλλαγή επήλθε απότομα. Η διαφοροποίηση είναι καλή γιατί οι λιγοστοί πόροι κατευθύνονται εκεί που υπάρχουν οι πραγματικές, οι αληθινές ανάγκες φτώχειας και μετά υπάρχουν τοπικοί πόροι διαθέσιμοι στις φτωχές χώρες. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση λέει ότι η διαφοροποίηση είναι καλή επιλογή. Όμως υποτιμήσαμε την περιπλοκότητα των καταστάσεων, την ποικιλομορφία τους, και το σημείο όπου κόψαμε ας πούμε τον αμφάλιο λόρο ήταν κάπως προβληματικό. Το σημείο που είπαμε ότι τώρα αποφυτίσατε και δεν χρειάζεστε κάτι άλλο. Υπάρχει και το θέμα της κινητοποίησης των εγχώριων πόρων, του να μπορούν να κινητοποιηθούν. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή, δηλαδή χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία, το Πακιστάν, ε, αν δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν επαρκώς τον τομέα υγείας ή παιδείας τους, όχι γιατί δεν δίδεται αρκετή αναπτυξιακή ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά γιατί δεν κινητοποιούνται επαρκώς διαθέσιμοι υφιστάμενοι εγχώροι πόροι. Και εμείς δίνουμε τέτοιου είδους πλαισίωση για να κινητοποιηθούν οι τοπικοί πόροι και να αντισταθμίσουν την έλλειψη εξωτερικής βοήθειας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ευθύνη αυτών των χωρών. Δεν μπορούν εύκολα να παρακάμψουν αυτό το ενδεχόμενο. Πρέπει να λειτουργήσουν και έτσι, αν όχι για να μειωθεί η φτώχεια, αλλά για να επιτευχθούν και άλλοι στόχοι για την ε, ε, αηφόρο ανάπτυξη Το CSO και τα LA προγράμματα του μέσω αναπτυξιακής συνεργασίας συνεχίζουν να αξιοποιούνται για αυτές τις χώρες. Αλλά και το GBGC, το Global Public Goods and Challenges, συνεχίζει να χρησιμοποιείται. Και υπάρχει και ένα άλλο εργαλείο που δεν ξέρουν πολλοί, που είναι χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Είναι το εργαλείο για την εταιρική σχέση και μπορεί και αυτό να αξιοποιηθεί σε αυτές τις χώρες. Εν πάση περιπτώσει, η αξιολόγηση συμπεραίνει ότι αυτές οι εναλλακτικέ δεν καλύπτουν όλα τα κενά 100%. Δεν θα πρέπει να έχουμε αδιαφοροποιητή προσέγγιση, να συνεχίσουμε να δίδουμε βοήθεια σε χώρες που έχουν επαρκείς εγχώριους πόρους από τη μία Άρα το ζήτημα είναι ακαθόδες, θα επανέλθω στο μέλλον, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας προσπαθεί να πλοηγηθεί σε ήρεμα νερά μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Αλλά σίγουρα κάτι λείπει, πρέπει να βρούμε τη λύπη, δεν είναι λύση να αναδιπλωθούμε στην προτέρα κατάσταση και στα προηγούμενα εργαλεία. Κυρία Πρόεδρε, Επίσης να πω το εξής. Από την έκθεση τα δύο πιο σημαντικά συμπεράσματα για τις μελλοντικέ προκλήσεις έχουν καταρχάς να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, με τα δικαιώματα για το φύλλο. Ένα από τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την έκθεση είναι ότι είναι όλο και πιο δύσκολο όλα αυτά να μπουν σε mainstreaming, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να πούμε ότι κάτι πρέπει να κάνετε για αυτά. Μας απαντάνε όχι. Τέλος σε πάρα πολλές χώρες ΑΚΕ αλλά και σε χώρες που ενεργοποιείται το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας μας απαντούν όχι με τίποτα τελειώσαμε. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργήσει μια κάποια μόχλευση όλων αυτών και να ασκήσει πίεση και άρα επιστρέφει στο βασικό ευρωπαϊκό εργαλείο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι σημαντικό. Και τι κάνουμε. Είναι απορία, δεν έχει λυθεί στο μέλλον. και πώς εξυγχρονίζει ε, εργαλεία η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει το SDG Agenda, το, το οποίο δεν βασίζεται σε δωρητές και λήπτες, αλλά σε διαπραγμάτευση, σε αποκοινού απόφαση, ε, σε πολλά και διαφορετικά πράγματα που δεν ταιριάζουν με το, την παραδοσιακή μακροπρόθεσμη συνεργασία. Δηλαδή, ε, όλη αυτή η συνεργασία γίνεται για άλλους σκοπούς και με άλλο τρόπο. Πώς όλα αυτά λοιπόν θα βρουν τη θέση που τους ταιριάζει εντός των εργαλείων, των μηχανισμών και των μέσων μας, αυτό είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση. Το Global Public Goods and Challenges είναι ένα σχετικά μικρό πρόγραμμα που προσπαθεί να κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα. Δεν ξεκινά εκ του μηδενός, αλλά είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση γιατί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε πλέον ένας μεγάλος ε, δωρητής, αλλά ένας συμμετέχον σε μια ευρύτερη ατζέντα όπου έχουμε συνεργάτες και αποφασίσουμε από κοινού. Όλο και περισσότερες ε, χώρες, ε, αν θέλετε, υιοθετούν μια κατηγορηματική στάση και μας λένε μας συγχωρείτε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι θέμα δικής μας πολιτικής και η πολιτική μας είναι ως εξής. Απέχει, χύψη. Και όλα αυτά πρέπει κανείς να τα έχει υπόψη του. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Θα ήταν ενδιαφέρον κάποια στιγμή να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε τι γίνεται με ε, ποια είναι τα διαφορετικά με το Global Public Goods and Challenges. Μας δώσετε κάποια στιγμή κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε τις προκλήσεις, όχι σήμερα, κάποια, κάποια άλλη στιγμή. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι μια νέα μορφή συνεργασίας. Δουλεύουν σε παγκόσμιο επίπεδο συνολικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης. Εκεί αποφασίζουν τα πράγματα, αλλά τελικά σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζονται στην πράξη. Έχουμε πολλά εργαλεία που προβλέπουν δηλαδή τη μελλοντική μορφή που θα πάρει η συνεργασία μας. Η Πρόεδρος. Και για το διάλογο με άλλους εταίρους πλην ε, κρατών, αυτό είναι πολύπλοκο και πολύπλοκο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όταν προσπαθούσα σε μία ε, περιφέρεια προσπαθώντας να δώσουμε κάποιο λόγο στους πολίτες επιτόπου για τα διαφορετικά ταμεία ε, είδα τις τεράστιες δυσκολίες ακόμη και πανεπιστημιακοί γράφουν βιβλία για το θέμα αυτό για αυτούς που υπεραμείνονται των συμφερόντων από όλες τις μεριές και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προβλήματα τα τα κράτη-μέλη δρούν συγκεντρωτικά σε επίπεδο κυβέρνησης και υπάρχει μία αντιπαράθεση με τις τοπικές αρχές και περιφέρειες. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση, όχι μόνο στα θέματα συνεργασίας με άλλες χώρες, αλλά και μέσα στις δικές μας χώρες. Μπορεί στην Ισπανία με τις αυτόνομε περιφέρειε να είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση, αλλά παραμένει η ένταση στο πώς λειτουργούν αυτά τα θέματα. Και είναι πολύπλοκο όταν μιλάμε για συνεργασία με χώρε όπου υπάρχουν δυσκολίε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά έχουν ε, καλύτερη απόδοση όσον αφορά την χρήση των αναπτυξιακών μέσων. Είναι θέματα για τα οποία δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, ευχαριστώ και την Επιτροπή που ήρθε στην, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε στην Επιτροπή μας. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα θέματα της αξιολόγησης. Ευχαριστούμε. Okay, colleagues, we're going to move on because we have... Ας συνεχίσουμε λοιπόν, συνάδελφοι, γιατί έχουμε περισσότερα σημεία. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 10, Παγκόσμια Πλατφόρμα για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, μια διάσκεψη που έγινε στο Κανκούν, στο Μεξικό, το Μάιο που μας πέρασε. Ο κ. Ε, Γκερέρο ήταν εκεί με τον Επίτροπο Στυλιανίδη και μπορεί να μας περιγράψει τι έγινε και τι θα είναι τα επόμενα βήματα. Ενρίκε. Ε, Ευχαριστώ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι στις 5 και 10 το απόγευμα πράγματι είναι απερίγραπτος ο ενθουσιασμός με τον οποίο η σεπτή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιμένει την έκθεσή μου για τα τεκτενόμενα στη Κανκούν στα τέλη Μαΐου. Προλίγου είχα λάβει πρόσκληση από πλευράς του Επιτρόπου στη Λιανίδη να αποτελέσω μέρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη συνεδρίαση που γινόταν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στη συνεδρίαση των συντονιστών της Επιτροπής Ανάπτυξης. Στη συνεστρίαση αυτή μάλλον αποφασίστηκε να υπάρξει αντιπροσωπεία ενός ατόμου, παρόλο που δεν συνηθίζεται για τέτοιου είδους ε, συνεδριάσεις. Οι συντονιστές όμως ε, αποφάσισαν αυτό δεν είναι μόνο προσωπική ενός προσώπου, γιατί και ο Μανουέλ Μανρίκε είναι πρόσωπο, είναι άτομο, άρα είχαμε διτή παρουσία και οι δυο μας πήγαμε και συνεδριάσαμε στην Κανκούν. Και πέρα από τις φωτογραφίες που βλέπετε στην έκδοση, ε, και σε μερικές από αυτές εμφανιζόμαστε με t-shirt, με κοντά μανίκια, να ξέρετε ότι καθόλου δεν πήγαμε για να αναψυχεί και ούτε αναψυχθήκαμε γιατί δεν μπορέσαμε καθόλου να βγούμε ε, η αίθουσα της συνεδρίασης ε, δεν είχε πρόσβαση στην ε, παραλία γιατί υπήρχε μια, υπήρχαν λόφοι από φύκια που εμπόδιζαν την πρόσβασή μας στο νερό. Και γι' αυτό δουλέψαμε εντατικά και δεν βγήκαμε από τους τέσσερις τείχους του, της αίθουσας όπου έγινε η συνεδρίαση. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη συνεδρίαση της συνολικής πλατφόρμας που έγινε μετά τη συνεδρίαση της ΕΝΤΑΗ πριν από δύο χρόνια, όπου και εκπονήθηκε και καταρτίστηκε το περιβόητο μάρκο του Σεντάι για τη μείωση των κινδύνων ε, καταστροφών με ορίζοντα τότε 2015-2030, ε, τη 15 ετία αυτή. Η Επιτροπή Ανάπτυξης απέστειλε αντιπροσωπεία και στο Σεντάι, πάλι με τον υποφαινόμενο και τον κύριο Ζέλερ μεταξύ άλλων, Έκτοτε άλλαξε από το Σεντάι στην Κανκούν η προοπτική του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές και με τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τον, τον αγώνα μας. Δηλαδή, εστρέψαμε το ενδιαφέρον μας όχι στην αντιμετώπιση, αλλά στην πρόληψη. Να είμαστε προετοιμασμένοι όταν συμβαίνουν και ε, λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Και έγινε συνεδρίαση στη Κανκούν δύο χρόνια μετά για να σημειώσουμε τι λειτουργήσε και τι δεν λειτουργήσε. Λοιπόν, Το σύνολο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν υπό την καθοδήγηση του Επιτρόπου Στυλιανίδη και η συνολική αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ της οποίας ήμουνα και εγώ μέλος, συμμετείχαμε σε διάφορες συνεδριάσεις με συνομιλητές από την Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών, από μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ. κτλ. Προσωπικά συμμετείχα σε συνεδριάσεις που είχαν πολύ πιο συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή το κοινοβουλευτικό σκέλος. Είχαμε για παράδειγμα συνεδρίαση μελών του Κοινοβουλίου που είχε οργανώσει η Γερουσία του Μεξικού και υπήρξε και εκεί παρέστηκε ο πρόεδρος της Ένωσης, Παγκόσμιας Ένωσης Κοινοβουλίων και μιλήσαμε για τις δράσεις των κοινοβουλίων και τη συνεισφορά τους στις στρατηγικές προετοιμασίας ε, και απάντησης και ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια ε, τέτοιου είδους κρίσεων. Επίσης συμμετείχα στην συνεδρίαση του Φόρουμ ΑΚΕ. Φόρουμ ΑΚΕ όπου παρέστησαν εκπρόσωποι από διάφορες χώρες και τόνισαν την ανάγκη οι περιφερειακές οργανώσεις να λειτουργούν και πώς οι περιφερειακές οργανώσεις πρέπει να ε, συστήνονται και να καθορίζουν γραμμές δράσης, να δίνουν κατευθύνσεις, κατευθυντήριες γραμμές, ώστε εκ των υστέρων όλα αυτά να ανεβαίνουν σε, σε περιφερειακό επίπεδο, σε κεντρικό επίπεδο, αλλά να κατεβαίνουν και σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στοιχείο κλειδί στρατηγικής σημασίας είναι η προετοιμασία των τοπικών αρχών για να υπάρξει έγκαιρη απάντηση στην κρίση. Από εκεί και πέρα συμμετείχα σε συνεδριάσεις ε, συνοδεύοντας όλη την υπόλοιπη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεδριάσεις όπου αναθεωρήθηκε η θέση που θα παρουσίαζε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Σύνοδο της Ολομέλειας, μέσα από την παρέμβαση του Επιτρόπου στη Λιανίδη. Δηλαδή συνεδριάσαμε για να διαμορφώσουμε το κείμενο της παρέμβασής του. Και ε, παρέστην και σε συνεδριάσεις με εκπροσώπους των ΜΚΟ και το εκπροσώπους οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, παρουσία του Γιωχάννες Λούχνερ που είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία του καθ' όλη τη διάρκεια της ε, παρουσίας μας και της παραμονής μας στην Κανκούν. Συζητήσαμε με τις ΜΚΟ, ε, είχαμε συζητήσεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες Μιλούμε για μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης για να ανταποκριθούμε έγκαιρα στις κρίσεις και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημάναμε ότι βεβαίως τυπικά υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε ε, την πυρίτιδα, αλλά πρέπει όλοι να συνειδητοποιούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πυροδοτηθούν αυτοί οι μηχανισμοί, να τεθούν σε λειτουργία. Και Κάποιος θα πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο να ε, ενεργοποιήσει το μηχανισμό. Αλλά γνωρίζουμε περί ποιου μηχανισμού πρόκειται. Αυτό δεν χρειάζεται καθόλου ψάξιμο πια. Και σημαντικό είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Είναι μια γενικότερη παρατήρηση αυτή σε πολλές περιπτώσεις και συχνά για την πρόληψη ε, από τις φυσικές καταστροφές είναι πολύ σημαντικό όλος αυτός ο κλάδος των ασφαλιών. Μιλούμε για εταιρείε ή για φορείς που μπορεί να είναι οντότητες νομικές δημόσιες, που μπορεί να είναι ιδιωτικές νομικές οντότητες και δίνουν δυνατότητα ε, ε, σε αντασφάλιση και σε κάλυψη άλλων ε, νομικών προσώπων που πλήττονται από παρατεταμένη ξηρασία, από περιπτώσεις επανειλημμένων πλημμυρών και το καθεξής. Και πρέπει εκεί να αναπτυχθεί και το δυναμικό και οι δυνατότητες των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των ΣΤΙΤ. προέκυψαν δύο έγγραφα στο τέλος, ανακοίνωση υψηλού επίπεδου, που υιοθέτησαν οι ηγέτες, η πολιτική ηγεσία για την διασφάλιση της ανθεκτικότητας και αντιοχής των υποδομών ε, και της ε, στέγασης. Υπήρξε επίσης ένα έγγραφο με την περίληψη, της σύνοψη ε, του Προέδρου, όπου γινόταν ένα είδος απολογισμού για το τι σημαίνει αυτή η παγκόσμια πλατφόρμα. Στη συνεδρίαση 7.000 άνθρωποι συμμετείχαν και περίπου 300 οργανώσεις. Τέλος, αυτή η συμμετοχή στην παγκόσμια πλατφόρμα και η συμμετοχή της δικής μας Επιτροπής στη συνεδρίαση του Σεντάι πριν από δύο χρόνια είναι οι βάσεις για να ενισχυθεί η θέση της Επιτροπής μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά και να συμβάλλουμε περισσότερο στο σχέδιο δράσης. Και αυτό το είδαμε και στη συζήτηση που είχαμε με τον Εστονό Υπουργό για το πρόγραμμα εργασιών της Εσθονικής Προεδρίας και Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει αυτό το έγγραφο το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου, αλλά και εγώ έχω εφιστήσει την προσοχή του Εσθονού Υπουργού στην ανάγκη και στην υποχρέωση τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να δρομολογούν και να εφαρμόζουν και να υλοποιούν σιγά-σιγά αυτό για το οποίο δεσμεύτηκαν σε διεθνή φόρουμ. Δεν είναι άλλωστε μόνο αποκλειστικά και μόνο δικός μας ο ρόλος εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά είναι και ρόλος των κρατών μελών να ε, κάνουν το παν για να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις και να υπάρξει πρόληψη. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες, η πρόληψη ε, συνεπάγεται τρομακτική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, αλλά και τρομακτική διάσωση ανθρωπίνων ζωών. Αυτό είναι κάτι που κατηγορηματικά αποδεικνύουν όλες οι διαθέσιμες μελέτες και πρέπει όλοι να το έχουμε υπόψη. Ευχαριστώ όλοι. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λίχνερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις για τον Ενρίκε. Έχετε κάτι να προσθέσετε για το ποια συνέχεια θα δοθεί σε αυτά. Θα είμαι σύντομος. Έχω τρία μόνο να παρατηρήσω. Πρόκειται για αυτήν την παγκόσμια πλατφόρμα που ήταν η πρώτη ευκαιρία ούτως ώστε να αξιολογήσουμε και να εφαρμόσουμε ε, το πλαίσιο του ΣΕΝΤΑ για την προσωπία της ε, Ένωσης με επικεφαλή στον κύριο Στυλιανίδη συμμετέχει σε πάνω από 30 εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, διμερείς συναντήσεις και ως επιτοπλίστων μέσα σε 48 ώρες επιβεβαιώνω όσα είπε ο κύριος Γκερέρο ούτε λεπτό για να πάει κανείς στην πλάζ. Οπότε και γι' αυτό και από τον ΟΗΕ και από όλους εμπλεκομένους είχαμε ε, συνοήσεις, ιδίως όσον αφορά πρακτικά θέματα της δουλειάς μας, η νομοθεσία για πολιτική προστασία, για ετοιμότητα, για πρόληψη, ε, δράσεις για τη μείωση του κίνδυνου, ε, χρηματοδότηση από τα ανθρωπιστικά ταμεία μας και επίσης ε, συστήσαμε και για επιστημονική έρευνα οπότε το θέμα ήταν συγκεκριμένο να διαπιστώσουμε ότι κάποιες χώρες όπως η Γουατεμάλα αναδέχθηκαν το δικό μας πλαίσιο για την μείωση του κινδύνου και τώρα το εφαρμόζουν σε όλη τους τη χώρα και ταυτόχρονα έχουν διαμορφώσει τη δική τους πολιτική πολιτικής προστασίας σε σχέση με αυτή την μεθοδολογία εμείς είχαμε την δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπήσαμε ε, στην, στο Τράπεζα την Υπουργική και στην ε, Τράπεζα Κορυφής. Επίσης ε, υπήρξε διμερές ενδιαφέρον έντονο κυρίως από τη Λατινική Αμερική. Κυβερνήσεις, εκπρόσωποι περιφερειών όπως το Μερκοσούρ και ζήτησαν να αντιγράψουν το δικό μας μοντέλο που είναι δύσκολο να γίνει απουσία εσωτερικής αγοράς, αλλά υπήρξε έντονο ενδιαφέρον όσον αφορά τις παρεμβάσεις της ε, σε Εκουαδόρ, Χιλή, Περού, Αϊτή. Ε, και πάλι αποδείχθηκε ότι είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στο έργο μας, οπότε και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον να αντιγραφεί το τι κάνουμε εμείς, γιατί θεωρήθηκε ότι αποτελεί προστιθέμενη αξία. Τέλος να σας πω ότι ένα από τα αξιοσημείωτα κατά τη γνώμη μου αλλά και κατά τη γνώμη του Επιτρόπου ότι λέω από την πρώτη συνάντηση η αντιπροσωπεία μας είχε συγκεκριμένη μενία θέση για στρατηγική για όλη τη διαδικασία και ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο με ΜΚΟ Οπότε και εκεί είχαμε το ίδιο μήκος κύματος. Ταυτότητα απόψεων, κρατή μέλη, κοινοβούλιο και κομισιόν, με μία φωνή. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για όλα όσα μας είπατε. Και τώρα περιμένουμε πώς και πώς τους καρπούς του έργου σας για να δούμε τι θα γίνει με τις καταστροφές και να έχουμε καλύτερο σύντονισμό. Και τώρα συνάδελφοι πάμε στο 11. Το τελευταίο για σήμερα. Το τελευταίο πριν τις διακοπές. Πολύ σημαντικό. Το τελευταίο, αλλά είμαστε ακόμα εδώ αρκετοί να συζητήσουμε τι γίνεται με τη στρατηγική με την Αφρική. Όθηση για ανάπτυξη. Έχουμε τώρα έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας Η συγητής μας είναι ο κύριος Μωρίς Πόγκα. Και θα κάνουμε τώρα, εν ώψη της του Αμπιτζάν, 29 και 30 Νοεμβρίου. Και είπαμε ότι εκεί θα είναι βασικό θέμα τι θα κάνουμε με τους νέους. Θα μια όδηση σχέση με την Αφρική και είπαμε ότι συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις κοινωνίες και απασχόληση για τους νέους και χτες βράδυ έβλεπα στην τηλεόραση ρεπορτάζ που έδειχναν βάρκες με νέους Αφρικανούς που ερχόντουσαν στην Ευρώπη και είμαι σίγουρος ότι όλες τις οικονομίες τις δώσανε στους λαθροδιακινητές ελπίζοντας να βρουν μια καλύτερη ζωή στην ε, Αφρική γιατί δεν υπάρχει καμία ελπίδα στη χώρα τους. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε. Κάτι καλύτερο να φτιάξουμε, να τους δώσουμε κάποια ελπίδα. Γιατί πολλές φορές κουβαλούν μαζί και την οικογένειά τους. Άρα κάτι πήγε το να αναλάβουμε δράση. Ο κύριος Πόγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας παρουσιάσω σύντομα το σχέδιο έκθεσης για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική. Μια όθηση για την ανάπτυξη. Είχαμε μια κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής ε, και της ΥΠΑ της Εκπροσώπου από τις 4 Μαΐου και θέλουμε να εκφράσουμε τις ε, προτεραιότητές μας ε, πριν την επόμενη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής που θα γίνει στο Αμπιτζάν 29 και 30 Νοεμβρίου του 2017. Αυτή η κοινή διακήρυξη είναι σημαντική και συμφωνώ με τα όσα προτάθηκαν και συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε την εταιρική μας σχέση με την Αφρική, που είναι μία ήπειρος με την οποία έχουμε στενές και προνομιούχες σχέσεις σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, αλλά και για την ανάπτυξη, την αναπτυξιακή, η ανθρωπιστική βοήθεια. Και είναι απόλυτα ε, σημαντικό να αναπτύξουμε τη σχέση μας με την Αφρική για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το σχέδιο έκθεσης έχει τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα τονίζω την αναγκαιότητα να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής για να ανανεώσουμε την εταιρική μας σχέση. Χρειαζόμαστε μια εταιρική σχέση από την οποία θα βγαίνουμε όλοι οι νικητές, θα βασίζεται στις δεσμεύσεις μας και στις ε, στρατηγικές που είχαμε μέχρι τώρα και που θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις που έχουν και οι δύο ήπειροι και κυρίως οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καλή διακυβέρνηση, μετανάστευση και περιβάλλον. Πρέπει να επανεξετάσουμε το πλαίσιο σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής και του αντίστοιχους δεσμούς και παράλληλα είναι σημαντικό να μην αμφισβητήσουμε το πλαίσιο χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακολουθήσουν άλλες ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ. Σύμφωνα με ε, τη συμφωνία του Κοτονού έχουν γίνει σημαντικές ε, πρόοδοι και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Ακόμη θέλω να τονίσω το ρόλο όλων των φορέων στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με την Αφρική θεσμική συνεργασία, αλλά και ρόλους της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα, ούτω ώστε η εταιρική σχέση να είναι ως το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και των δύο υπήρων. Το δεύτερο τμήμα του σχεδίου έκθεσης αφορά το θέμα της ανθεκτικότητας και του ρόλου των νέων που θα αποτελέσει βασικό ζήτημα στην ε, συνάντηση του Νοεμβρίου. Πρέπει να μιλήσουμε για την ανθεκτικότητα σε όλες τις, τις διαστάσεις. Καταρχήν, πολιτική ανθεκτικότητα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη χρηστή διακυβέρνηση και να τονίσουμε τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους συναδέλφους μας στην Αφρική και θα πρέπει να δηλώσουμε εκ νέου ότι η αναπτυξιακή βοήθεια έχει ως προϋπόθεση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την χρηστή διακυβέρνηση. Δεύτερον, ανθεκτικότητα στον τομέα της ασφάλειας. Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια και αντιστρόφως. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της Αφρικής σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας και ε, οι αφρικανικές χώρες θα πρέπει όλο και περισσότερο να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους θέματα. Επόμενο θέμα, η ανθεκτικότητα στον τομέα του περιβάλλοντος. Η Αφρική πλήθεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και αποτελεί δική μας ευθύνη να υπενθυμίσουμε τις δεσμεύσεις του Παρισίου και να υποστηρίξουμε διάφορες πρωτοβουλίες ούτως ώστε το εμπόριο φυσικών πόρων να είναι περισσότερο διαφανές. Υποστηρίζω μια χάρτα Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Τέταρτον, ανθεκτικότητα στον οικονομικό τομέα θέλω να τονίσω τον καθοριστικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ε, που θα επιτρέψει τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα στις χώρες της Αφρικής. Ακόμη, το θέμα της δημιουργίας μιας ζώνης ε, ελευθέρων συναλλαγών στην Αφρική και συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Όσον αφορά την κοινωνική ανθεκτικότητα, είναι σημαντικά τα θέματα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της υγείας. Αυτά αποτελούν προτεραιότητα και πρέπει να δίδονται ευκαιρίες στους νέους, διαφορετικά δεν θα θέλουν οι νέοι να παραμείνουν στην Αφρική. Το τρίτο τμήμα του σχεδίου εκθέσεως αφορά την κινητικότητα και τη μετανάστευση. Έχουμε εκπονήσει πολλές εκθέσεις για αυτά τα θέματα. Δεν προσπαθούμε να είμαστε ε, πλήρεις, αλλά θέλουμε να τονίσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα για τις σχέσεις μας με την Αφρική. Τονίζω τη σημασία που έχει μια συντονισμένη προσέγγιση ε, στα θέματα της κινητικότητας και της μετανάστευσης και να προσπαθήσουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για αυτά τα θέματα ανάπτυξης της Αφρικής. Θα πρέπει να είναι επιλογή η κινητικότητα και η μετανάστευση και να μην είναι κάτι το οποίο υφίσταται ο πληθυσμός. Δεν μπόρεσα να είμαι ε, απόλυτα λεπτομερής ε, για όλα τα θέματα, αλλά νομίζω ότι οι συνάδελφοι και σκιώδεις συζητητές θα εμπλουτίσουν το σχέδιο έκθεσης με τις παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Ήδη ε, έχουν ζήσει το λόγο κάποιοι συνάδελφοι και δίνω το λόγο στο Νόβερτ Νόιζα. Ευχαριστούμε, Μωρίς. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό το σχέδιο έκθεσης. Και ελπίζουμε ότι στην ε, συνάντηση στην ακτή του Ελεφαντοστού θα συζητηθεί λεπτομερέστερα και θα ε, εγκριθεί. Μας απασχολούν θέματα όπως η καταπολέμηση της ε, φτώχειας και το θεματολόγιο του 2030 και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν συνένεση από αυτού. Και θα πρέπει και το πλέγμα κινητικότητα και μετανάστευση να εξεταστεί σε αυτό το πνεύμα. Η Ερυθρέα που συζητήσαμε το πρωί αποτελεί ένα παράδειγμα. Αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία αποτελεσματική παρακολούθηση θα πρέπει να είναι προϋπόθεση. Μπορεί να περνάμε μέσα από καταπιστευματικά ταμεία για τη δημιουργία ε, ε, ανάπτυξης ε, επιτόπου. Αυτά θα αποτελέσουν τη βάση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Για τη μετανάστευση, στο τελευταίο κομμάτι του σχεδίου έκθεσης, εκεί όπου αναφέρεται η μετανάστευση και η κινητικότητα, θέλω να πω ότι είναι σημαντικό θέμα, αλλά και αμφιλεγόμενο. Είναι μια πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα πρέπει να επισκιάζει τους μακροπρόθεσμους στόχους της Επιτροπής μας. Θα πρότεινα μια κάπως διαφορετική διατύπωση λοιπόν στο τελευταίο αυτό κομμάτι της έκθεσης το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο που είναι εταίρος μας θα πρέπει επίσης να τονιστεί όπως και ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζει. Η ανάπτυξη και τα αναπτυξιακά μέσα πρέπει να αποτελέσουν ε, ένα σημαντικό μέσο να προωθήσουμε τις επενδύσεις που θα βοηθήσουν ε, τους μικρούς γεωργούς και τις οικογένειες, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας, θα πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση στο νερό, τα δικαιώματα στις χρήσεις γης, ε, και την, τα δικαιώματα στη χρήση σπόρων. μέσω ε, πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προωθηθούν οι επενδύσεις με την τήρηση των κανόνων ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για θέσεις απασχόλησης που θα σέβονται την αξιοπρέπεια η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση για όλους θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα διασφαλίσουμε, ιδίως για τους νέους, καθώς ε, και ε, ικανοποιητικές συνθήκες υγείας. Αυτά ε, θα ενδυναμώσουν τις χώρες της Αφρικής και τμήμα της στρατηγικής μας θα πρέπει να είναι και το θέμα της δημογραφικής αλλαγής. είναι μια τεράστια πρόκληση. Βλέποντας την, Ιγερή, την Ιγυρία, για παράδειγμα, που σε λιγότερο από μία γενιά μπορεί να έχει τριπλασιαστεί ο πληθυσμός της, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και συμφωνώ με τον Μωρίς Πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της συμφωνίας ε, του Κοτονού. Αυτά τα οποία κάνουμε εδώ με αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά με ε, τη συμφωνία του Κοτονού. Ευχαριστώ. Judith Sargentini. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και συνάδελφε Πονγκά. Η προπαρασκευή για το Αμπιτζάν μας κάνει να πρέπει να προσέξουμε περισσότερο την Αφρικανική Ένωση. Σε σχέση με αυτό που συζητούμε σήμερα, ξέρω ότι οι πράσινοι θέλουν να αντιταχθούν στην παράταση της ε, Κότονου. Αν θέλουμε να χειραφετήσουμε την Αφρικανική Ένωση θα πρέπει όλα αυτά να τα θεωρήσουμε ενιαίο θέμα και έτσι να το προσεγγίσουμε. Όχι όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει κάνει αυτούς τους διαχωρισμούς. Πού δηλαδή υπάρχει θέμα μετανάστευση που δεν υπάρχει. Νομίζω δεν βοήθησε την προσέγγιση μας στη συνάντηση κορυφής της Βαλέτας. Πρέπει τα αφρικανικά θέματα να τα προσεγγίζουμε όλα μαζί. Να μην έχουμε αυτό το σκοτεινό σύννεφο πάνω από την Αφρική. Θα πρέπει να τα δούμε με υγιή τρόπο τα ζητήματα στο Αμπιτζάν. Εμείς θεωρούμε ότι τα θέματα του Αμπιτζάν θα πρέπει να μην σχετίζονται με μετανάστευση και Ευρώπη. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια στην Ευρώπη, αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να μην ανακατεύουμε τα ζητήματα των αιτίων και αιτιών της μετανάστευσης. Άρα, σε αυτή την έκθεση, Μωρίς, θα πρέπει να τονίσουμε το πώς θα αντιμετωπιστεί η ανισότητα πώς θα πρέπει η προσοχή μας και η χρηματοδότησή μας να πάει στην Αφρική για την καταπολέμηση της φτώχειας με βιώσιμο τρόπο και καταπολέμηση και των ανισοτήτων. Σήμερα κιόλας είχαμε δύο ομάδες εργασίας. Για την Ερυθρέα τα είπαμε εδώ, για τη χρηματοδότηση και στις 1.30 είχαμε άλλη ομάδα εργασίας και εξετάσαμε τα προγράμματα για τον Νίγηρα μέσω του Αφρικανικού καταπιστεύματος. Θα πρέπει, είπαμε, για τον Νίγηρα να καταπολεμηθεί η λαθρομετανάστευση. Δεν έχει τρόπο χρηματοδότησης ο κόσμος. Και ο κόσμος για να βρει χρήματα γίνεται διακινητής μεταναστών. Δεν είναι σωστό δεν είναι βιώσιμο. Θα πρέπει να δούμε ότι έτσι υπάρχει περισσότερη ανασφάλεια. Όλα είναι και περισσότεροι πεθαίνουν τώρα στο Νίγηρα γιατί τους εγκαταλείπουν στην έρημο. Βλέπουμε περισσότερους νέους χωρίς δουλειά. Και εκεί αυτοί αυτομάτως έχουν περισσότερη ανασφάλεια. Από πού προέρχεται η ανασφάλεια. Αυτό να δούμε πολλές φορές είναι για πολλούς νέους που δεν έχουν κάτι να κάνουν στην ε, ζωή. Δεν έχουν σαν στόχο να φροντίσουν η οικογένεια. Αυτά επικρίνουμε. Και επίσης αυτό το οποίο δεν καλύπτεται από το σχέδιο κειμένου, είναι, δεν είναι απαντήσει σε πολλά. Αλλά πρώτα πρώτα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κοινή ανακοίνωση για μια νέα όθηση στην εταιρική σχέση Ευρώπης-Αφρικής. Γίνεται μια πλημνία, αλλά όχι με λεπτομέρειες. Επίσης, θα θέλαμε να δούμε στην έκθεση κάτι άλλο. Τη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας εταιρική σχέση. Θα πρέπει να αξιολογηθεί αν τα πράγματα έχουν τη σωστή κατεύθυνση. Άλλο που αναφέρεις, αλλά θα μπορούσαμε να το βελτιώσουμε, για το τι γίνεται με την φοροδιαφυγή. Τα λες εκεί ξεκάθαρα, αναφέρεις τα 50 δις δολάρια ετησίως, τα οποία φεύγουν από την Αφρική γιατί δεν καταβάλλονται σχετική φόρη γι' αυτό είναι πολύ επιζημίο για αναπτυσσόμενες χώρες. Ξέρετε ότι τώρα έχουμε την Ερευνητική Επιτροπή για την φοροδιαφυγή, για τα Panama Papers. Άρα θα πρέπει αυτό να τα πούμε. Θα βοηθήσει αυτό για τη συνάντηση του Αμπιτζάν και αυτό θα βγάλει κάτι. Παίρνουμε χρήματα από την ανάπτυξη και τα πάμε στην μετανάστευση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αρέσει στους από την Αφρική. Τέλος τα προγράμματα κινητικότητα. Η μετανάστευση φυσικά και θα συζητηθεί στο Αμπιτζάν, αλλά σας παρακαλώ μπορούμε να μιλήσουμε και για τις δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης. Φοιτητές, εργαζόμενοι, να κάνουν κάτι χρήσιμο στην Ευρώπη, να φέρουν τις δεξιότητές τους. Και κατόπιν να δούμε το θέμα της ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι επομένω η έκθεση αυτή προωθεί τη συνεργασία. Θα πρέπει εμεί να δώσουμε απαντήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Um, Dziękuję bardzo, <clears throat> panie Przewodnicząca. E, chciałem pogratulować i e, serdecznie podziękować. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Πόγκο για αυτό το σχέδιο έκθεση. και να συγχαρώ και όλους τους συναδέλφους που έχουν ήδη συμμετάσχει και που θα συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της έκθεσης αυτής. Η έκθεση αυτή αφορά το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο παγκόσμιος πολιτισμός. Όταν συζητάμε τέτοια θέματα, ακούγεται συχνά η άποψη ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τους φτωχούς. Θέλουν ε, οι πλούσιες χώρες να βοηθήσουν τις φτωχές χώρες. Μία λοιπόν ε, ε, προσέγγιση πλούσιων έναντι φτωχών χωρών. Εγώ πιστεύω ότι εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια διάσταση και είναι ένα πρόβλημα που έχει σχέση με τον πολιτισμό μας. Ο σημερινός μας κόσμος είναι ένας κόσμος όπου η ζωή διαδραματίζεται γρήγορα. Θέλω να πω με αυτό ότι οι κοινωνικές διαδικασίες διαδραματίζονται τόσο γρήγορα, περνάνε μπροστά από τα μάτια μας ε, μέσα σε λίγα χρόνια και όχι σε διάστημα γενεών όπως γινόταν παλιότερα. Γιατί σας έκανα αυτή την εισαγωγή. Εκτιμώ ιδιαίτερα την δουλειά του κυρίου Πόγκα και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα καθήκοντα. Πρώτον, θα πρέπει να δράσει περισσότερο στεναρά σε ένα παγκόσμιο συνασπισμό μεταξύ κρατών του Βορρά παγκοσμίω για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Αφρικανικής Υπήρου. Δεύτερον, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική με κάποιους ακρογωνιαίους λίθους, με κάποιους στόχους που θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Μέχρι τώρα ακολουθούσαμε μία συγκεκριμένη προσέγγιση, δηλαδή ανθρωπιστική βοήθεια, ε, φιλανθρωπική δράση. Υποστηρίζουμε με τη δράση μας τους πλουσίους της Αφρικής, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο διαφθοράς και κλιματικής δραστηριότητας στην Αφρική. Βλέπουμε ότι αν μεταφέρουμε χρήματα χωρίς συγκεκριμένε προϋποθέσεις δεν θα φτάσουν στην τσέπη εκείνων που θα θέλαμε να υποφεληθούν από την αναπτυξιακή βοήθεια. Οποιαδήποτε λοιπόν βοήθεια δίδεται θα πρέπει να δίδεται υπό όρους, να είναι συγχρηματοδοτούμενη μεταξύ χωρών δωρητών και χωρών που λαμβάνουν τη βοήθεια και θα πρέπει να τίθενται και ορισμένες προθεσμίες για την επίτευξη στόχων. Αν αυτοί οι όροι δεν πληρούνται, θα πρέπει να μην παράσχεται η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν θα πρέπει να συνεχίζεται να χορηγείτε ή και να αποσύρετε. Δεν είναι Βαρέλη, δίχως πάτο η Αφρική. Είναι σημαντική η βοήθεια για όλους τους λαούς, σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να δώσουμε άλλα 40-50 χρόνια, άλλες 2-3 γενιές. Δεν έχουμε το χρόνο για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Γιατί όπως σας είπα, στην τωρινή κατάσταση λίγα χρόνια έχουν αντικαταστήσει τι γενιές ή τους αιώνες του παρελθόντος. θέτουμε το πλαίσιο με διάφορες ιδέες και στη συνέχεια αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βάλει το σωστό περιεχόμενο. Αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε συγκεκριμένα κριτήρια για το πώς θα αποκομίσουμε αυτά τα οποία θέλουμε, με τι όρους, μέσα σε τι χρονικά πλαίσια και με ποιες συγκεκριμένες δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σεσίλ Κιέγγε. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λίντα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Μωρίς για την ε, έκθεση που μας παρουσίασε ξεκινά ξανά η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο υπήρων, της Ευρωπαϊκής και της Αφρικανικής Υπήρου. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η αναπτυξιακή βοήθεια, η βοήθεια για τη δημιουργία νόμιμων οδών μετανάστευσης αναδεικνύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι παράγοντες. Και ένα βασικό στοιχείο που έλειπε, το υπογράμμασα στην πρώτη μου παρέμβαση, είναι ο ρόλος της διασποράς. Οπότε άφησαν την Ήπειρό τους και έχουν συμβάλει στις οικονομίες της χώρας προέλευσης. Και λέμε θα πρέπει να ξαναχαρακτηθούν κάποιες πολιτικές. Πολλές κοινωνικές πολιτικές αφρικανικών χωρών ενισχύονται από αυτά τα εμβάσματα. Αυτά τα εμβάσματα που είναι πιο μεγάλα ποσά από οποιαδήποτε άλλη βοήθεια προς την ε, Αφρική. Άρα θα πρέπει, είπαμε, να κοιτάξουμε και το θέμα της διασποράς. Συμβάλλουν πολύ τα εμβάσματα στην οικονομία πολλών χωρών. Και όπως έλεγα προηγουμένως, είναι σημαντικό αυτό να ενισχύσουμε αυτό που είπε ο Νόρμπερτ, να δούμε δηλαδή τι θα γίνει για την περίοδο μετά την Κοτονού. Να ληφθεί και αυτό η υπόψη και να χαραχθεί μια στρατηγική γι' αυτό στα πλαίσια της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης με την Αφρική. Να υπάρχει μια προσέγγιση από την οποία όλοι να βγουν κερδισμένοι. Είναι σημαντικά αυτά που λέει ο Μωρίς. Θα πρέπει και δύο πλευρές να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους μέσα από μια τέτοια εταιρική σχέση. Να θεωρήσουμε ότι δεν είναι μόνο Αφρική και Ευρώπη τώρα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Σε αυτή τη λογική να μπούμε. Αυτή τη λογική να υιοθετήσουμε να ενισχύσουμε τις χώρες με διάφορες χώρες, πολιτικά και οικονομικά. Ακριβώς όπως τα λέει η έκθεση, ανθρωπικότητα, αντοχή. τελευταία αποστολή που κάνουμε στην Αφρική μας έδειξε ότι όλοι λένε εκεί δεν βλέπουμε πού είναι οι επιπτώσεις, πού είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών των πόρων που πάνε εκεί. Πολλές χώρες και πολλοί που ήταν δικαιούχοι της ε, βοήθειας κατήντησαν να εξαρτώνται από την οπτικσιακή βοήθεια. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε τα μέσα τα οποία οδηγούν σε ανθεκτικότητα τον πληθυσμό και εν κατακλείδη θέλω να σας πω ότι θέλω να αναλάβω την έκθεση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που αφορά την κινητικότητα και την μετανάστευση. Και θέλω σε αυτή την εκθεσή μου να αναφέρω κάποια στοιχεία που δεν τα βρήκα εδώ στο τμήμα του κειμένου που λέει για την ε, μετανάστευση και την κινητικότητα. Εγώ θα προσπαθήσω αυτά τα θέματα να τα αναδείξω στην ε, έκθεση που θα συντάξω. Και ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε. Σισίλια. Ο κύριος Βέντα. Και εγώ να ευχαριστώ τον κύριο Πονγκά για τη δουλειά του. Πολύ σημαντικό το θέμα. Είναι η έκθεση, τονίζει πολλά θέματα και τονίζει το ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των πολιτικών και συντονισμός Ένωσης και κρατών μελών. Όπως είπατε, τονίζεται αυτές τις πέντε διαστάσεις της ανθεκτικότητας ολοκληρωμένη προσέγγιση χρειάζεται. Να μην βλέπουμε απομονωμένους τομείς. Τον δυτικό τομέα και τις πολιτικές που εφαρμόζουν τις δράσεις που φροντίζουν την ανθρώπινη ασφάλεια με παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών. Uh, Εγώ πρόεδρε να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Η μετανάστευση παραμένει σημαντικό στοιχείο των σχέσεών μας με την Αφρική. Να αλλάξει το αφήγημα. Ανάπτυξη και μετανάστευση να τα δούμε σε σχέση με τον στόχο των στατικών υπαριθμών 10. Έχουμε IP, ε, τα πιστεύματα, όλα αυτά είναι μέσα χρηματοδότησης. Αλλά πρέπει να κανονίσουμε όλα αυτά να καταφέρονται κατά της φτώχειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Μην περιοριζόμαστε σε ελέγχους συνοριακούς. Η ελευθερία διακίνησης είναι κάτι πολύ βασικό. Είναι κάτι για το οποίο υπερηφανευόμαστε. Γιατί να το υπονομεύουμε στην Αφρική. Και σήμερα όπως ελέγχθη είχαμε αυτή την ε, ομάδα εργασία. Ε, εντυπωσιάζει το πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε τη δουλειά μας. Όπω όπως είπε η κυρία Σαρτζεντίνη, είδατε τι αντίκτυπο είχαν τα, η δουλειά μας στο στον Νίγηρα. Υπάρχουν ε, θέματα και στο της μετανάστευσης. Τώρα ήδη αναφέρθηκε το θέμα της ε, φορολογίας. Τα τελευταία 50 χρόνια είπαμε ότι υπάρχει απώλεια ενός 3 δολαρίων. Άρα θα πρέπει να επιμείνουμε, θα πρέπει η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή να καταπολεμηθούν στην Αφρική. Εδώ υπάρχει αυτή η, η για το δημοκρατικό μέρισμα. υγεία αναφέρεται μόνο μία φορά στην έκθεση. Μπορούμε να πούμε περισσότερα. Να διαπιστώσουμε ότι θα πρέπει να προσεχθεί περισσότερο το θέμα των ασθενειών στην Αφρική. Κοινωνική σημασία, της πρόσβασης σε γενετήσια υγεία και αναπορικά δικαιώματα. Να πρέπει να πετύχουμε τους στρατηγικούς στόχους, να βελτιώσουμε το επαγγελματικό περιβάλλον με περισσότερη αναπτυξιακή συνεργασία. Ευχαριστούμε τον Σιγητή και τους Σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω δύο δικά μου σχόλια να κάνω. Και στη συνέχεια είχα προσχεθεί στον Λουί Μισελ να του δώσω το λόγο να διαβάσει μία δήλωση από ένα συνάδελφο της ομάδας του. Αλλά είναι στα γαλλικά και μου ζήτησαν να το διαβάσω εγώ αντί για τον αντιπρόεδρο. Θα το διαβάσω εντός λίγο. Όμως έχω να πω δύο πράγματα δικά μου. Πρώτον, για τα φορολογικά συμφωνώ με την κυρία Σαρτζεντίνη. Πριν από λίγα χρόνια συναντήσαμε το Θάμπο Μπέκι Μιλήσαμε για τη συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση. Μας είχε ζητήσει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με αυτή την Ένωση και νομίζω ότι η Επιτροπή θα μας μιλήσει για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης, να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση, κάτι να κάνουμε. Να δούμε ποια συνέχεια δόθηκε στη σχετική έκθεση, να συνεργαστούμε με τον εισηγητή. Αυτό καταρχάς. Δεύτερο, για την κοινωνική ανθεκτικότητα για τους νέους. Να γίνει ειδική μνήμα στη στήριξη των νέων γυναικών. Δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων στην Αφρική αν δεν αλλάξουμε τις ζωές των νέων γυναικών, να έχουν επιλογές, να έχουν μέλλον. Άρα να μιλήσουμε για τη διάσταση του φίλου. Έγινε εξαιρετική συνεδρίαση και διάσκεψη πριν από λίγες εβδομάδες. Έγινε λόγος για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για την υποχρέωση παροχής εκπαίδευσης και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Και θα ήθελα τώρα να διαβάσω τη δήλωση του Λουί Μισελ, που είναι σκιώδης εισηγητής για το Άλντε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τον Μωρίς Πονγκά για την εξαιρετική του έκθεση για τη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική. Δεν έχω πολλά να προσθέσω παρά μόνο το γεγονός ότι στην επόμενη σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής, Αφρικανικής Ένωσης, η Ένωση Αφρικανικών κρατών που θα γίνει στην Αμπιτζάν το Νοέμβριο του 2017 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στρατηγικές προοπτικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα της εταιρική σχέσης για να έχουμε και σωστή συνοχή μεταξύ ε, της διαδικασίας μετά το Κοτονού και της εταιρικής σχέσης ΕΕ χωρών Αφρικανικών Αφρικανικής Ενότητας. Ο περιφερειακός πυλώνας είναι κάτι που θα εξεταστεί στην Αμπιτζάν. Με άλλα λόγια, η προτεραιότητά μας θα ενταχθούν στο πλαίσιο της ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας μετά τη διαδικασία του Κοτονού. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής για να γίνει η πραγματικότητα υπό τον όρο ότι θα έχουμε ισότιμη διανομή του πλούτου που θα δημιουργείται. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε την εκ νέου απίκηση και απεικιοκρατική κατάκτηση, αν θέλετε, της Αφρικής. Καλό όλους να ενταχθούν και να συμμετάσχουν σε αυτό το πολιτικό διάλογο για να αντιμετωπίσουν τα διακύβευματα, τα μεγάλα της εποχής μας και να μιλήσουμε με μια φωνή ενιαία στα διεθνή φόρουμ. Οι χώρες ΑΚΕ είναι το 40% των μελών, χωρών μελών των, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα ήθελα να σας το επιθυμίσω για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν είχε να μας πει ο Λουί Μισελ για τη διαδικασία μετά το Κοτονού, να μιλήσουμε όλοι με μια φωνή στα Διεθνή Φόρουμ, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην παρουσιάζεται διαιρεμένη. Να καλέσω τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράση να μας πούν δύο λόγια. Ο κύριο Ντομένικο Ρώσο πρώτα και η κυρία Χαβά στη συνέχεια. Ντομένικο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Λίντα, που μου δίνει το λόγο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Φτάνει σε κατάλληλη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κατά την προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής στα τέλη Νοεμβρίου. Πρέπει, όπως πολλοί ομιλητές τόνισαν, να τονίσουμε την γεωπολιτική σημασία της Αφρικής Θυμίζω ότι η Αφρική και η Αφρική είναι ο πρώτος μας, ε, μάλλον η Ευρώπη ο πρώτος εταίρος για την Αφρική και για το εμπόριο και για την ανάπτυξιακή βοήθεια και η διάσκεψη κορυφής στο Αμπιτζάν είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε για να δηλώσουμε εκ νέου τη σημασία αυτής της εταιρική σχέση και για να οικοδομήσουμε αυτή την εταιρική σχέση πάνω σε καινούρια βάση. Υπάρχουν και νέοι φορείς ε, στο παιχνίδι, αλλά είναι σαφές το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να παραμείνουμε η πρώτη εταίροι της Αφρικανικής Υπήρου. Φέτος λοιπόν έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή για να δημιουργήσουμε μια σωστά προσανατολισμένη εταιρική σχέση. Ακόμη και αν αυτή η ευκαιρία απαιτεί μια τεράστια επένδυση, όχι μόνο χρηματοοικονομική, αλλά και πολιτική επένδυση. Και το τόνισαν αυτό πολλοί ε, βουλευτές που έλαβαν το λόγο. Πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι το 2035 η Αφρική πρέπει να δημιουργήσει τουλάχιστον 8 ε, εκατομμύρια νέε θέσει εργασία και αυτέ οι νέε θέσει εργασία πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια των αξιοπρεπών θέσεων εργασία, όπω είπατε πολλοί από εσά. Λαμβάνοντα υπόψη τη σχέση τις ε, σχέσεις μας με την Αφρική και τις συμφωνίες μετά το Κοτονού δεν υπάρχει καμία ε, αντίφαση. Είναι συμπληρωματικές αυτές οι δύο δυναμικές και αλληλοενισχύονται. Και θέλω να ε, πω ότι την περασμένη εβδομάδα έγινε μια πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση για να προετοιμάσουμε τη συνάντηση με την Αφρικανική Ένωση και η Αφρικανική πλευρά πρότεινε να δοθεί η ονομασία Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρικανική Ένωση. Μπορεί να είναι η πέμπτη διάσκεψη κορυφής που οργανώνουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Αφρική, αλλά θα είναι η πρώτη διάσκεψη κορυφής που θα αποκαλείται διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης και αυτό το ζήτησε η Αφρικανική πλευρά. Και δεν θα πρέπει να πούμε όχι σε αυτό το αίτημα της αφρικανικής πλευράς. Νομίζω ότι συμφωνούμε λοιπόν για τους στόχους και για την προοπτική αυτής της διάσκεψης κορυφής και νομίζω ότι η έκθεση αυτή και το ψήφισμα που θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα δράσουν συμπληρωματικά και θα ενισχύσουν αυτή τη συνιστόσα, δηλαδή όχι μόνο αναπτυξιακή σχέση αλλά και πολιτική σχέση μια εταιρική σχέση που συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα των σχέσεων με την Αφρική. Η Αφρική είναι η πιο κοντινή μας Ήπειρος, είναι μια Ήπειρος που η δημογραφία της δημιουργεί προβλήματα αλλά και ευκαιρίες για την Ευρώπη, για το μέλλον. Όπως είπα λοιπόν πριν, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να μας ξεφύγει. Και αυτό θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να τονίσει ιδιαίτερα η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Χέν Χαβας, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ, Λίντα. Τα είπε όλοι ο Ντομινίκα, αλλά να συμπληρώσω κι εγώ δύο σχόλια υποστηρίζουμε την έκθεση και συγχαίρουμε τον εισηγητή για την ε, ε, προσέγγιση του. Και συγχαίρω και το Κοινοβούλιο για την συμμετοχή που έχει σε αυτή τη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Αφρικής. Μια μικρή πρόταση, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά τον τίτλο να λέμε εταιρική σχέση και όχι στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής, γιατί δεν είναι μια νέα στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόγκα, θέλεις να απαντήσεις ε, στους συναδέλφους Μωρίς. Απλώς να ευχαριστήσω, Πρόεδρε, τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο για τις παρατηρήσεις τους και ανυπόμονα περιμένω τις τροπολογίες τους. Θεωρώ ότι ομονοούμε για τα θέματα της ε, έκθεσης. Περιμένω τις τροπολογίες σας και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν. Σας θυμίζω ότι η προθεσμία είναι συνάδελφοι πρώτη ενάτου στις 11 η ώρα για τις τροπολογίες. Ε, άρα γιατί όλο το καλοκαίρι να φτιάξετε τις τροπολογίες. Μπα, καλύτερα κάντε το τώρα πριν φύγετε και τα ξεχάσουμε όλοι. Έχουμε δύο θέματα. Δώδεκα. Ωραία ρωτήσουν, Δεν υπάρχουν ρωτήσεις. Δεκατρία. Διάφορα. Όχι. 38 στις εννέα. Και το απόγευμα την επομένη. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Καλή ξεκούραση στις θερινές διακοπές. Μια που όλοι σκληρά εργαστήκαμε και αξίζουμε τις διακοπές μας.